Είναι Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξή σας έχει αποσταλεί. Το έχετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Να θυμίσω ότι τα σημεία 10, 11 και 12 τη ημερήσια διάταξης, δηλαδή όσο έχουν να κάνουν με την τροποποίηση του κανονισμού, του δημοσιονομικού κανονισμού που θαρμάζεται για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τις ευρωπαϊκές κοινότητε, με εισηγητή τον κύριο Ριβελίνη, θα τα δούμε από την Επιτροπή Προπολογισμών στις 17.45 αύριο, 6 παρατέταρτο δηλαδή. 6 παρατέταρτο με 6.30. Την απόφαση αυτή την λάβαμε στη διάσκεψη των ε, Προέδρων την περασμένη 8 Ιουλίου και βάσει του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου με το και βάσει του άρθρου 54 θα γίνει κοινή εξέταση από τις δύο επιτροπές των νομοτήσεων αυτών. Έγκριση των πρακτικών στο σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης πρακτικά της συνεδρίασης της 26 η και 27 η Απριλίου 2010 και της 21ης Μαΐου 1 η Ιουνίου 2010. Έχουν αποσταλεί από την 5η Ιουλίου. Ως, ε, όπως και άλλες φορές μπορείτε, η συνεδρίαση μας μεταδίδεται και στο διαδίκτυο και βλέπετε ότι προβλέπονται ψηφοφορίες για τα σημεία 4 και 5 της ημερήσιας διάταξη. οπότε θα ψηφίσουμε με την κάρτα μας ηλεκτρονικά. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4. Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Μαρινέσκου. Ο συνάδελφο Μαρινέσκο είναι στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου θα ήθελα και εγώ να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, λέει η κυρία Γκρέσλε. Αλλά τι να κάνουμε. Ε, για την ψηφοφορία δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο. Έχουμε συζητήσει και με τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Μια προφορική μονοτροπολογία θα ήθελα να υποβάλω στην τροπολογία υπαριθμών 14, όπου την εποπτεία θα την κάνουμε έλεγχο. Το supervision να γίνει scrutiny στα αγγλικά. Έτσι, όχι supervision εποπτεία, αλλά scrutiny, έλεγχος. Κατά τα άλλα νομίζω είναι σημαντικό ε, στις τροποποιήσεις του οργανισμούς να είμαστε σοβαροί και υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αφορούν όλους τους οργανισμούς αυτούς ε, επί της αρχής. Και έτσι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να βελτιώσουν και τη λειτουργία τους γενικά και μεγαλύτερη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Είναι το πρώτο βήμα πραγματικά σοβαρής ε, αντιμετώπισης και βελτίωσης των προβλημάτων και των ελλημάτων που είδαμε και στην έκθεση Ματιού. Αυτά τα ολίγα και τελείωσα. Ε, Ευχαριστούμε, συνάδελφε Γκρέσλε. Εάν όλοι έχετε λοιπόν τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, να περάσουμε στην ψηφοφορία για το σημείο 4. Ψηφίζουμε λοιπόν. Voto per alzare di mano. Voto manuale. Manual vote. Ok. Allora, poniamo in Θα ψηφίσουμε λοιπόν την τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να ψηφίσουμε ομού τις τροπολογίες σαν μπλοκ. Ας εκφραστούν και οι άλλες πολιτικές ομάδες. Εμείς παντού έχουμε θετικό πρόσημο, ορισμένοι άλλοι έχουν αρνητικό. Μέχρι το πρώτο αρνητικό δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Διαφωνείτε με την αμπλοκ ε, ε, ψηφοφορία όλων των ε, τροπολογιών. Dann stimmt einfach mit uns. Τότε ψηφίστε τη δική μας λίστα. Ja, die ersten drei. Οι τρεις πρώτες. Μέχρι και την τρία. 26, 1, 2, 3. Αυτές τις τέσσερις δεν μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί όλες. Την τέταρτη χωριστά και μετά θα ξαναπροσπαθήσω να ζητήσω on μπλοκ. Forse facevamo prima se proseguiamo. Comunque. Ίσως να έπρεπε αυτό είχαμε κάνει, αλλά θα είχαμε ήδη τελειώσει. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, από κοινού τι τέσσερι πρώτε 26, 1, 2 και 3. Άρχεται η ψηφοφορία. La Πέρας. Εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία περιθμών 4, άρχεται η ψηφοφορία. Votazione Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε συνολικά τις τροπολογίες από 28 έως 30, έως και 30. Σωστά. Ε, ε, ε. Όχι, υπάρχει αντίρρηση. Οπότε ψηφίζουμε μία προς μία. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα Εγκρίνεται. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Με την προφορική της τροπολογία. Πέρας. Εγκρίνεται. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το τελικό σχέδιο γνωδότησης, όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Τέλεια. Συνεχίζουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Σημείο 5. Εδώ και πάλι προβλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίου έρευνας. Το λόγο για κύριο Πατρικέλο. Πρόεδρε, δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω. Επί του θέματος, περαιτέρω προφορικές τροπολογίες δεν υπάρχουν και συμφωνούμε με το σχέδιο γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε. Περνούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Έτοιμοι. Τροπολογία πρώτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Θέλετε να ψηφίσουμε on block, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ναι. Από την 1 έω την 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνονται με 21 ψήφου υπέρ, 1 κατά και ψηφίζουμε το τελικό σχέδιο γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Ευχαριστώ. Eh, Και τώρα ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 6. Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με, τα, τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμηση τη Απάτης, Όλαφ. Εδώ θα έχουμε παρουσίαση από τον Επίτροπο υπεύθυνο για την ε, καταπολέμηση της απάτης και, τη φορολογική, και το φορολογικό έλεγχο, τον κύριο Σέμετα. Εξαφανίστηκε όμως ο Επίτροπος. Non c'è. E che vogliamo fare? Andiamo avanti. Facciamo l'otto. Non c'è. Allora, siccome il commissario... Il commissario... Επειδή ο Επίτροπο Σεμέτα δεν είναι ακόμα εδώ και για να μην χάνουμε χρόνο, επειδή είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διαταξή μα με πολλά θέματα, να περάσουμε στο σημείο 8, διότι το 7 σημείο θα το δούμε τελείως μετά το 9ο, την, ε, το θέμα της κυρίας Ματιέ. Να δούμε τώρα το θέμα του κυρίου Μπαλτσίτη στο σημείο 8, το σύνολο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έφτασε. Ε, έφτασε ε. ο Επίτροπος, τον βρήκανε. Έρχεται. Σε μετά ή Βαλτσίτης, γιατί είμαστε Λιθουανοί και οι δύο. να περάσουμε τώρα στην αρχική σειρά της ημερήσιας διάταξη. Έφτασε ο Επίτροπος Σεμέτα, τον ευχαριστώ και του δίνω το λόγο για να μα παρουσιάσει το έγγραφο το σχετικό με την Όλαφ. Παρακαλώ. Alla parola, commissario. Prego. Distinguished members, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία μου εδώ για να σας παρουσιάσω αυτό το έγγραφο για, τις, για τη λειτουργία της Όλαφ και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που μπορέσαμε να το ετοιμάσουμε πριν τας διακοπάς. Έχει υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και το θεωρώ τεράστιας σημασίας για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε την μεταρρύθμιση της λειτουργίας της ολαφ και ειμαι ιδιαιτερα ικανοποιημένο που μπορεσαμε να το ετοιμασουμε πριν τα διακοπας εχει υποβληθει στο ευρωπαικο κοινοβουλιο και το συμβουλιο και το θεωρω τεράστια σημασιας για να δουμε πως θα συνεχισουμε την μεταρρυθμιση τη λειτουργιας της ολαφ Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα του φορολογουμένου και της φορολογουμένης θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση των απατών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν η Όλαφ να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να καταπολεμήσει την διαφθορά, απάτη ή οτιδήποτε άλλο απειλεί τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Έχουμε αναλάβει την κοινή δέσμευση να είναι υπόλογη πλήρωση Όλαφ και να σέβεται ταυτόχρονα, να σέβονται και οι άλλοι ταυτόχρονα την πλήρη της ανεξαρτησία. Μπορεί να έχουν τεθεί ερωτήματα, τίθεται μάλλον το ερώτημα πώς θα το πετύχουμε αυτό. Εμείς ταυτίσαμε συγκλίνοντα και αποκλίνοντα θέματα στις θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη σύγκριση, σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής του 2006 για να δείτε και εσείς πώς μπορείτε να καταλήξετε σε καλύτερη συμφωνία. Όλες οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Κομισιόν συνεργάστηκαν για τη σύνταξη του εγγράφου μας και το έγγραφο έχει την εξής δομή. Πρώτον, θέματα που έθιξαν τα άλλα όργανα τα περισσότερα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Μερικά είναι ακόμη εκκρεμή. Η προσθήκη 1 περιγράφει τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις για τα προβλήματα αυτά, τονίζοντας ιδιαίτερα που υπάρχει σαφής διαφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Η προσθήκη 2 έχει έναν πίνακα με τις θέσεις των τριών οργάνων και με παραπομπή στον σημείο του εγγράφου όπου αναφέρεται η διαφωνία. Το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η συγγήτρια κυρία Γκλέσλερ έκαναν πολύτιμη συμβολή και τόνισαν ορισμένα σημεία δικαιότατα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Όλαφ. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την κυρία Γκρέσλερ για τις προσπάθειές της να βελτιώσει την Όλαφ. Κοίταξα προσεκτικά όλα τα θέματα που έθιξε το ψήφισμα του ΕΛΚ του Νοεμβρίου, του Κοινοβουλίου με συγχωρείτε, και μερικά πρόσθετα θέματα. Μερικά από αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά όπως η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των προσώπων που την χάνουν έρευνας και ιδιαίτερα έρευνας από την όλαυση σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα, σώματα και υπηρεσίες καθώς και με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ο ορισμός γενικού διευθυντή της έρευνας και μιας επιτροπής που να την παρακολουθεί. τα θέματα που μας χωρίζουν αφορούν την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Όλαφ, τη διάρκεια των ερευνών αυτών, βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Όλαφ και οργάνων της Ένωσης καθώς και Όλαφ και κρατικών αρχών, καθώς και με την Ευρωπόλ, την Ευρωτζάστ και τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Εδώ τίθεται και το θέμα του ρόλου του διευθυντή της Όλαφ. Η πολιτική διακυβέρνηση σημαίνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Όλαφ και άλλων σωμάτων, δημόσια πληροφόρηση από την Όλαφ, σεβασμό των δικαιωμάτων των ερευνουμένων κλπ. Για όλα αυτά τα θέματα έχω υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις που μπορεί να αποτελέσουν λύσεις στα θέματα που μας χωρίζουν. Στην προσθήκη 1 θα τα βρείτε αυτά. Παραδείγματο χάρη, η Επιτηρητική Επιτροπή της Όλαφ δεν θα παριορίζεται στο να παρατηρεί κατά πόσον γίνονται σεβαστοί οι κανόνες που διέπουν τις σχέσεις με τα άλλα όργανα, αλλά και την εξέλιξη των ερευνών και πρέπει επίσης η Επιτροπή αυτή να μπορεί να κάνει και συστάσεις για την, για την ε, ταύτιση των προτεραιοτήτων της όλα αυτής διαρκείας των ερευνών της και του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμόζονται οι συστάσεις που αναφέρει το εγχειρίδιο της Όλαφ. Προσεχώς, προσεχώς. Τώρα, νομίζω ότι Δύο είναι τα κύρια προβλήματα ή προκλήσεις. Πρώτον, να βρεθεί κατάληξη ισορρόπηση μεταξύ ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας της Όλαφ και ευξημένη υπολογισμότητά της μάλλον. Να είναι υπόλογη δηλαδή η Όλαφ. Η συνεργασία μεταξύ Όλαφ και άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης και σωμάτων και υπηρεσιών καθώς και κρατών μελών πρέπει να γίνει με τέτοιο και αυξημένη υπολογισμοτητα ώστε να συμβαδίζει με τις πρακτικές απαιτήσεις της έρευνας, της κάθε έρευνας. Οι προελίσεις που προτείνουμε λοιπόν πρέπει να αφήνουν χώρο σε κάποια ευελιξία που να επιτρέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ερευνών και να συμβάλλει στην μικρότερη διάρκεια τους. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να καθορίσουμε ρητά το ρόλο της Επιδυτικής Επιτροπής με τρόπο ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με κανένα άλλο όργανο υπηρεσία. Θα δείτε ότι ορισμένες λύσεις έχουν προταθεί και γι' αυτό και στο κυρίως κείμενο και στην πρώτη προσθήκη. Μερικά από τα θέματα εκκρεμούν ακόμη και άρα απαιτούν περαιτέρω συζήτηση. Όπως η καλύτερη λύση που πρέπει να βρεθεί μεταξύ του, για τον διάλογο μεταξύ οργάνων και πολιτικής διακυβέρνησης της Όλαφ. Επίσης πρέπει να δούμε αν άλλοι ενδιαφερόμενοι όπως η Ευρωάστ και η Ευρωδίκ δεν πρέπει να παίξουν και αυτές κάποιο ρόλο. Είμαι πεπισμένος ότι βάσει του εγγράφου αυτού μπορούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για να προχωρήσουμε και να βρούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Σας είχα παρουσιάσει πριν από ένα μήνα ένα έγγραφο για την απαλλαγή ως προς τις ε, έρευνες που έχουν γίνει ή θα γίνουν για τη δωροδοκία και τη διαφθορά και θα βρείτε και γι' αυτό ορισμένες προτάσεις στο έγγραφό μας. Μπορεί να έχετε δει ότι το έγγραφο προτείνει λύσεις με βάση όλες τις προτάσεις που έχει κάνει το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν βέβαια ακόμη ορισμένα σημεία επί των οποίων δεν έχουμε συμφωνήσει πλήρως, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές εναλλακτικέ λύσεις ώστε να μπορούμε να πούμε ότι θα βρεθεί και για αυτά λύση. Παραδείγματο χάρη, είναι ανάγκη όλες οι υποθέσεις να παραπέμπονται στα εθνικά δικαστήρια όπως προτείνει το Κοινοβούλιο. Υπολογίζω στην υποστήριξή σας και τις επόμενες εβδομάδες γιατί ο διάλογος αυτός θα καθοδηγήσει την Κομισιόν να υποβάλει μια τροποποιημένη πρόταση για τις έρευνες που διενεργεί η Όλαφ. Ελπίζω ειλικρινά η Κομισιόν να μπορέσει να κάνει αυτή την τροποποιημένη πρόταση πριν λήξει το έτος. Στόχος είναι να καταλήξει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι το 2011 και προσβλέπω σε καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, κυρία Γκρέσλε. Είναι καταπληκτική ημέρα σήμερα. Χριστούγεννα και Πάσχα την ίδια μέρα πέσανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ε, ε, τηρήσατε την υπόσχεσή σας. Πραγματικά για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό και πολύ ευίωνο. Την τελευταία εβδομάδα, την Τετάρτη μου δώσατε ένα έγγραφο. Το Σαββατοκύριακο δεν το κοίταξα σε μεγάλο βάθος, έτσι λίγο το ξεφύλισα. Χρειάζεται μεγάλη ανάλυση και επιμελή. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί πραγματικά είναι μια βάση για διαβούλευση. Και πήραμε από την αρχή μία περιστατωμένη έκδοση για να δούμε ε, πού υιοθετείτε τις απόψεις έκθεσης και πού όχι. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο Κοινοβούλιο είναι να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο έγγραφο που εμείς εγκρίναμε. Γιατί δεν είναι μόνο συντριπτική πλειοψηφία, περίπου 95% αλλά είναι και διακομματική. 92 τροπολογίες που σε μεγάλο βαθμό τις συνυπογράφουν κοινέ πρωτοβουλίες των πολιτικών ομάδων μετά από προτάσεις του εισηγητού. Δηλαδή δεν είναι ούτε έγγραφο του ΕΛΚ ούτε δικό μου, είναι πραγματικά κοινή δουλειά του Κοινοβουλίου. Και θα ήταν για μας σημαντικό όσο γίνεται ε, να υιοθετήσετε τις προτάσεις μας και με τη σειρά τις προτεραιότητές μας συμφωνούμε απολύτως νομίζω ότι σε πρώτο πλάνο θα πρέπει να βρίσκεται ο ρόλος των κρατών μελών. Δηλαδή, πώς συνεργάζονται με την Όλαφ, πώς συνεργάζεται η δικαιοσύνη, πώς τα διαβιβάζει αυτά και τι κάνουν οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τη στατιστική που έχω δει εγώ, Μόλις 7% των περιπτώσεων της Όλαφ καταλήγουν στη δικαιοσύνη και μάλιστα με δικαστική απόφαση, άρα το 93% καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Ε, αυτό πώς σας φέρετε; Όποιος έχει ακόμα μια στοιχειώδη πίστη και οι βουλευτές πρέπει να πιστεύουν στη δικαιοσύνη, αυτή η κατάσταση είναι αφόρητη. Γι' αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα και δική μας και θα πρέπει οπωσδήποτε το Συμβούλιο να ανταποκριθεί. Τώρα, πώς θα συνεργαστούμε εμείς για την καταπολέμηση της απάτης με το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό και ε, για πολύ καιρό επίμαχο, διαφωνούσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να πιέσουμε και χαίρομαι που βλέπετε με καλό μάτι την πρότασή μας. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία όπου μια φορά το χρόνο να συνεδριάζουμε μαζί με το Συμβούλιο. Όχι δηλαδή τι κάναμε τώρα, ότι συζητάμε με την Εποπτική Αρχή, με την αντίστοιχη Επιτροπή ε, και εκ του σύνεγέ συνομιλίας ο καθένας ξεχωριστά να τα λέει με την Όλαφ, ε, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, όχι, από κοινού να έχουμε μια κοινή πολιτική, να συζητούμε μια κοινή πολιτική και να την εφαρμόζουμε για την καταπολέμηση της απάτης και έτσι θα μπορούσαμε να προτείνουμε και πολλά για βελτίωση. Βλέπω λοιπόν ότι έχετε υλοποιήσει ε, τα όσα προτείναμε. Να με συμπαθάτε, δεν μπορώ, σας είπα, να μελετήσω και να αναλύσω το έγγραφο, δεν θα αναφερθώ σε όλα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ για το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια σημαντικά σημεία έχει κάνει κάποιες χαλαρωτικές, ας πούμε, κινήσεις. Ε, έχετε αποτινάξει την ιδεολογία που σας διείπε πριν από 1,5 χρόνο. Ο προκάτοχός σας, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να το πω, ναι. γιατί είναι σημαντικό για να βρούμε κοινέ λύσεις. Έχουμε κοινό συμφέρον, κοινέ λύσεις να βρούμε, να λειτουργήσει καλύτερα η Όλαφ από ό,τι μέχρι σήμερα. Αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν εδώ ιερές αγελάδες, ότι ε, αυτό το α, το β, το γ δεν το θίγουμε με τίποτα. Όχι. Και ο Review Advisor, ο αρμόδιος για τις διαδικασίες είναι ένα θέμα που το συζητάτε επίση. Διάφορε αλλακτικέ προτάσει. Επίση πολύ σημαντικό. Θα κοιτάξουμε τι προτάσει, θα μελετήσουμε ποια είναι η καλύτερη και σωστά παραπέμπεται εδώ στο εγχειρίδιο τη Όλαφ. Μήπω θα μπορούσε εκεί να λυθεί πώ συνδέεται ο Γενικό Διευθυντή σε μια ηγετική δομή στο εσωτερικό τη υπηρεσία. Δεν λέω ότι το βλέπω αρνητικά. Απλώ υπάρχουν σήμερα κάποια ε, προβλήματα, κάποιες αδυναμίες στον κανονισμό και αυτά περνάνε μέσα από το Γενικό Διευθυντή που έχει μια ιδιάζουσα και μοναδική θέση στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να το δούμε. Υπάρχει αυτή η ιδέα των checks and balances, δηλαδή να έχουμε εξουσίες και αντεξουσίες, βάρη και αντίβαρα. Ε, να το ξαναδούμε αυτό. Ε, θα Έλεγα λοιπόν ότι πρέπει από κοινού να πείσουμε το Συμβούλιο να ξανανοίξει το θέμα, να εκπονήσετε ένα νέο έγγραφο πραγματικό ουσιαστικό για τις διαβουλεύσεις και θέλουμε να πούμε και εμείς τη γνώμη μας, οι συντονιστές να συζητήσουν πώς θα το κάνουμε. Έκθεση πρωτοβουλίας, γρήγορα, έγγραφο εργασίας, δεν ξέρω τι μορφή θα λάβει, που να θεωρείται έκθεση πρωτοβουλίας και το έγγραφο εργασίας με τροπολογίες. Νομίζω αυτό είναι πιο ευέλικτη λύση θα το δούμε αυτό στην ομάδα εργασία και οι ηγητές ε, διακομματικά να αναλύσουμε και πάλι τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας και να σας κάνουμε προτάσεις τι μπορείτε να περιμένετε από εμά και τι όχι. Κατά τα άλλα δεν έχω ένα πρόβλημα εγώ και να συγκρουστώ και να διαπληκτιστώ με το Συμβούλιο και να διαφωνήσω. Ανησυχώ. Γιατί σε ό,τι αφορά τη Βελγική Προεδρία για το δημοσιονομικό κανονισμό δεν θέλει να κάνει τίποτα. Αυτό μου λένε οι επαφές μου. Και αφού αδράνησαν και οι προηγούμενες προεδρίες και ακολουθούν οι Ούγγροι και δεν θυμάμαι ποιο άλλο μετά και δεν θέλει να θίξει τίποτα, ε, κάτι πρέπει να σκεφτούμε κι εμεί. Μήπως στον προπολογισμό του 2011 να <laughs> προβλέψουμε καμιά έτσι δυσάρεστη ε, διάταξη για να τους τρομάξουμε. Είναι το σημαντικότερο αυτό και για μας και απέναντι στους πολίτες, άνδρες και γυναίκες που έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους σε εμά να βελτιώσουμε την κατάσταση και στην Όλαφ. Λοιπόν, και μια που καθόμαστε εδώ και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, τι γίνεται με το Γενικό Διευθυντή, ε, τρέχει η διαδικασία. Υποτίθεται ότι συμμετέχουμε κι εμείς και καλό θα ήταν να μάθουμε πώς θα συμμετέχουμε και πώς θα κινηθεί αυτή η διαδικασία για το διορισμό. Νομίζω ότι θα πρέπει το συντομότερο και μας ενδιαφέρει να αρχίσει να λειτουργεί ε, και να αναλάβει καθήκοντα. Σας ευχαριστώ ενδιαφέροντα αυτά που μας προτείνετε και σας ευχαριστώ επίσης που χαλαρώνετε λίγο τη θέση σας, ότι τηρήσατε το λόγο σας πραγματικά και ε, δεν τα κοιτάτε όλα αυτά με ιδεολογικές αγγυλώσεις. Και θα είμαστε πραγματικά στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ačiū gerimas e, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ θα επαναλάβω τις ευχαριστίες που εξέφρασε και συνάδελφος για την ετοιμασία αυτού του πολύπλοκου θέματος και εγγράφου και που το υποβάλλατε και εγκαίρο στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλο σας το έργο. Δεν θα περάσω σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει κανεί να έχει ιδιαίτερη πείρα σε αυτό το τομέα για να μπορεί να εκφραστεί με βεβαιότητα. Αλλά η Όλαφ, όπως και άλλοι θεσμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώ χρήζει μια μεταρρύθμισης έστω και εν μέρη. Θα συμφωνήσω λοιπόν με την κυρία Γκρέσλε ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν σοβαρέ ελλείψεις ισορροπία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλά από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Όλαφ αφορούν πολλές φορές και το ίδιο το κύρος των 27 κρατών μελών. Πρέπει να είμαστε ικανοί να αποδείξουμε ότι είναι χρηστή η αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο για την συνεργασία μεταξύ της Όλαφ και των αρχών των κρατών μελών, εδώ συμφωνώ με τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου ότι θα πρέπει οι εκθέσεις πρόοδου και τα προγράμματα πρόοδου, τα action plans, να υποβάλλονται από τα κάτι μέλη εγκαίρως. Θα πρέπει λοιπόν ενδεχομένως να μεταρρυθμίσουμε τις σχετικές διαδικασίες για να γίνουν ταχύτερες. Και όσο για τη συνεργασία τη Όλαφ με την Europol, τη Eurojust και άλλου διεθνεί οργανισμούς, είναι ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό δεν έχει φυγεί Ω τώρα αρκετά, δεν έχει συζητηθεί αρκετά. Είναι όμω αναγκαία μια τέτοιου είδου συνεργασία. Και αυτό θα πρέπει να το προβλέψουμε στο μέλλον. Για τι περιπτώσει απάτης που έχουν ε, αμελητέ επιπτώσει. θα συμφωνήσω με την άποψη ότι δεν θα έπρεπε εδώ να διαχωρίσουμε τι περιπτώσει ίσονο και μείζονο σημασία. Και όσο για την Επιτροπή Εποπτείας, Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο αν θέλουμε να παραμείνει όλα ανεξάρτητη και να καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα. Η λειτουργία αυτής της ε, Επιτροπής Εποπτείας θα πρέπει να ενισχυθεί και στο μέλλον. Και όσο για τους συμβούλους που ασχολούνται με συγκεκριμένε περιπτώσεις απάτης, είμαι προσφυγές από κράτη-μέλη, Νομίζω αυτή την αρμοδιότητα θα μπορούσε να την αναλάβει ακριβώς η Επιτροπή Εποπτείας. Να συμπεριλάβει δηλαδή αυτές τις θέσεις στην συνολική της δομή. Εάν δεν υπάρχουν απόρριτες πληροφορίες, εμπιστευτικέ, θα πρέπει να παραμένουν τέτοιες, δηλαδή απόρριτες. Αυτό δεν φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει πρόβλημα. Όσο για το διορισμό του Γενικού Διευθυντή, Νομίζω το πρόσωπο που θα, διορίζε, θα διορίζεται θα πρέπει να εργαστεί με τρόπο πιο ποιοτικό και να αποδείξει ότι είναι ικανό και για κάτι τέτοιο. Και όσο για τη διάρκεια της θητείας νομίζω ότι θα πρέπει να παραταθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα ε, της εργασίας του και της επιδόσης του. Σε ό,τι αφορά το θέμα των εντολών που θα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής, το θέμα είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Όμω, ο Διευθυντής θα πρέπει στο μέλλον να μπορεί να αποφασίζει ποιε είναι οι κύριε έρευνε και οι κύριε αρμοδιότητε που θα πρέπει να αναλαμβάνει, ανάλογα με την φύση τη κάθε έρευνα. Είναι πολλά όσα έχουμε να κάνουμε ακόμη σε αυτό το τομέα και συμφωνώ εδώ με την συνάδελφο. Θα πρέπει να συντάξουμε ένα έγγραφο όπου να καταγράφουμε συγκεκριμένε προτάσει και σχόλια, προσπαθώντα να βελτιώσουμε όχι μόνο το έργο τη Όλαφ, αλλά το έργο όλων μα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφο Γιάλα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάλα. Κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους μου για την παρουσίαση του κειμένου από τον Επίτροπο εντός του διαγράμματος. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε και εγώ δεν είχα χρόνο να τα μελετήσω. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αν μη τι άλλο θα ήθελα να αναφέρω αυτή τη στιγμή γιατί τα θεωρώ ουσιαστικότατα. Θα επιθυμούσα να σας ε, επενθυμίσω, επιτρέπετε ότι το Κοινοβούλιο επανειλημμένος έχει τονίσει και έχει απαιτήσει να υπάρξει και κώδικα συμπεριφοράς και δοντολογία σε περίπτωση σφαλμάτων που υπήρξαν στην Όλαφ να ε, βρίσκεται κάποια λύση. Βέβαια με τις δικονομικές εγγύησεις ε, των ε, ατόμων ή των οργανώσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση και ανάκριση. Όλα αυτά καλά και θα πρέπει να βγουν στο κείμενο. Και όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, αυτό ο επόπτης και η ε, επιτροπή που ελέγχει όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα τα ξαναδούμε, θα τα ξανασυζητήσουμε δεν ξέρω, σου φταίει το γεγονό ότι δεν είχα χρόνο να διαβάσω τα παραρτήματα. Πάντως στο κείμενό σας μιλάτε για την ανάγκη να αυξηθεί το έργο του, να έχει και άλλε υποχρεώσεις και καθήκοντα. Δεν διαφωνώ, αλλά σε καμία περίπτωση να μην περιορίζουν ε, τη δυνατότητα της Επιτροπής αυτής να ε, έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε ε, ενημέρωση. Μην τυχόν δηλαδή και περιορίσουμε αυτή την επιτροπή. Θέλουμε να είναι και ανεξάρτητη η Όλαφ, αλλά και ε, να διασφαλίζονται όλες οι δικονομικές εγγύσεις και τα διαδικαστικά θέματα. Και για τις σχέσεις με την Ευρωπόλ και Ευρωτζάστ, να μας πει ο Επίτροπος τι προβλέπεται εκεί, εάν θα έχουμε και προς τα εκεί μια πασαρέλα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, για αυτή την ε, υπόθεση που συζητούμε τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για πώς θα συνδεθεί η Όλαφ με αυτή την πορεία προς το μέλλον. Συμφωνώ και με τον κύριο Βαλτσίτης και με την κυρία Γκρέσλε για το θέμα του Γενικού Διευθυντού. Νομίζω ότι ορίστε αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της διαδοχής ή της εκλογής μετά από μια κατάσταση, πώς να πω, ε, αυτή τη δυστυχή έκφραση που είχαμε μετά την απώλεια του προηγουμένου διευθυντού και σε σχέση με τα κράτη-μέλη θα θέλαμε να ξέρουμε τι συνέχεια θα δίνεται, τι παρακολούθηση των διαδικασιών και πώς αυτά θα δημοσιοποιούνται στην κοινή γνώμη. Και όσο περισσότερα τα έχει έγκαια, τόσο καλύτερη η διαδικασία, πιο εύκολη και πιο ε, σωστή. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω, και να τονίσω πάλι αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλερ ο κύριος Έρενχάουζερ. Μόνο το 7% καταλήγει στα δικαστήρια. Αυτό μπορεί να είναι θέμα όπου να φταίει η εισαγγελία ή όλα η ίδια για τις μεθόδους που έχει, τις δυνατότητες διερεύνησης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πιστεύετε ότι φτάνουν μόνο τόσο λίγες υποθέσεις στο δικαστήριο. Ένα άλλο θέμα, μου επιτρέπετε σύντομα, είναι το σημείο 3. Ενημέρωση της κοινή γνώμης για τις έρευνες Σόλαφ. Στο παρελθόν επανειλημμένα είχαμε δει να γνώριζε ο τύπος νωρίτερα κάποια στοιχεία ή ποιος είναι υποδιερεύνηση πριν το γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το αντικείμενο ή το υποκείμενο της διερεύνησης. Υπάρχουν εσωτερικοί μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων. Μέχρι σήμερα εφαρμόζονται και ποια ε, προβλέπετε εξέλιξη για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε. Uh, thank you, Mr. Uh, Chairman. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, περισσότερο δηλώσεις έγιναν παρά ερωτήσεις, αλλά θα σας πω μερικά λόγια για το θέμα. Λοιπόν, πρώτον, δεν πρόκειται παρά για μια απλή παρουσίαση των αντιδράσεών μας προς τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Είναι πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα θα είναι μια πληρέστερη συζήτηση και των συγκεκριμένων επιλογών που έχουμε και που προτείνονται εδώ. Μπορώ απλώς να σας επιβεβαιώσω ότι τα θέματα που ενδιαφέρουν τους βουλευτές όπως οι σχέσεις Όλαφ και κρατών μελών, συμμετοχή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στη δραστηριότητα της Επιτηρητικής Επιτροπής, Εποπτικής Επιτροπής, Αυτά και άλλα θα καλυφθούν, καλύπτονται από το εγγραφό μας και προτείνονται και εναλλακτικέ λύσεις ως προς το πώς να τα χειριστούμε όλα αυτά και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι για ειλικρινή συζήτηση επί των προτάσεων αυτών αφού είναι κοινό ο στόχος μας. Να καταστήσουμε την Όλαφ εργαλείο αποτελεσματικό. Οι αριθμοί που ανέφερε η κυρία Γκρέσλερ, το 7% δηλαδή των ερευνών που παρακολουθούνται από τις χώρες μέλη μόνο 7%. Ο πραγματικός αριθμός είναι μάλλον υψηλότερος όταν αν σκεφτούμε το γεγονός ότι μερικές έρευνες χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλες. Δεν μπορούν όλες να συζητηθούν και να λυθούν αμέσως από το κράτος μέλος. Αλλά βέβαια το θέμα της διάρκειας μιας έρευνας είναι όντως ένα θέμα και θα θέσουμε πολύ συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια ώστε η Όλαφ να μπορέσει να, συντομεύει, να συντομεύσει τις έρευνές της. Και η Εποπτική Επιτροπή θα το κοιτάξει αυτό. Θα το κοιτάξει. Θα δει τι γίνεται με τις έρευνες και θα πρέπει η Όλαφ να μπορεί να εξηγεί κάθε φορά γιατί μία έρευνα χρειάζεται περισσότερο χρόνο από τους 12 μήνες που απαιτούνται τώρα ας πούμε στο εγγραφό μας. Για τη συνεργασία με την Ευρωάστ και την Ευρωδίκ επί προτείνουμε και επ' αυτού στο ίδιο το κείμενό μας του τροποποιημένου κανονισμού να υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια δηλαδή οποιοδήποτε ευρωπαϊκό σώμα ή οργανισμός να πρέπει να πρέπει να εφαρμόζει τη συνεργασία με την Όλαφ για την Ευρωάστη και την Ευρωδίκη συγκεκριμένα αυτές οι διατάξεις υπάρχουν ήδη, προβλέπονται. Η Όλαφ έχει ήδη συμφωνία με την Ευρωδίκ και για συνεργασία και με την Ευρωάστ γίνονται συνεννοήσεις. Εφόσον καταλήξουν αυτές θα δούμε τι θα λένε. Λοιπόν, για το ρόλο της Εποπτικής Επιτροπής στο έγγραφο βλέπετε ότι προτείνουμε σημαντική ενδυνάμωση της και βέβαια αυτή η Εποπτική Επιτροπή πρέπει και να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που χρειάζεται. Ούτως ή άλλως θα διασφαλίσουμε οι έρευνες καθεαυτές να, να ή μάλλον η πληροφόρηση επί των ερευνών καθεαυτών, καθεαυτών των design ερευνών να είναι πλήρης, πλήρης η πληροφόρηση και για να μην δημιουργούνται προβλήματα με την, σχετικά με την ανεξαρτησία της Όλαφ κατά τη διεξαγωγή των ερευνών. Αλλά, όπως σας είπα και πριν, προτείνονται εναλλακτικέ λύσεις στο έγγραφο. Μερικά ερωτήματα για την ισχύουσα διαδικασία ορισμού του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή της Όλαφ Μπορώ να σας πω απλώς ότι η διαδικασία ε, γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ακολουθείτε και παράλληλα στην Κομισιόν συζητιούνται τα πράγματα, αν και η Εποπτική Επιτροπή είναι, εργάζεται και αυτή σε όλη τη διαδικασία και η, ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι εκείνος που προτείνει ο οδικός χάρτης για τον ορισμό γενικών διευθυντών της 20 Σεπτεμβρίου αν δεν απατώμε φέτος, φέτος, φέτος, του, όχι ακόμα δηλαδή, οπότε και θα καθοριστούν οι υποψήφοι και θα αρχίσουν οι συνεντεύξεις και, και αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο οπότε και θα έχετε άμεσες επαφές με τους υποψηφίους για τη θέση του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ. Αυτά σύντομα είναι τα θέματα που τέθηκαν. Η κυρία Γκρέσλερ επίσης μίλησε και για προεδρίες Ε, και για την ομοθεσία εκεί της Όλαφ, ε, για τις προεδρίες, η Βελγική Προεδρία και οι επόμενες, η Ουγγρική και η Πολωνική, ναι, ε, πιστεύω ότι θα, θα κατορθώσουν να αρχίσουν τη συζήτηση αυτής της διαδικασίας τροποποίησης της νομοθεσίας μετά από συζητήσεις βέβαια με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά. Και η Κομισιόν τότε θα αρχίσει την καθεαυτού διαδικασία. The link of with uh, EPPO. E, e, e μετά κάποιος ρώτησε για το EPPO που λέμε. Το λέει το έγγραφο το ΙΠΠΟ, το γράφει για ΙΠΠΟ, κάτι λέμε εδώ στο έγγραφο. ΙΠΠΟ. Η διαδικασία, η διανομοθετική διαδικασία για την τροποποίηση της νομοθεσίας της Όλαφ θα καταλήξει σε μια πιο αποτελεσματική λειτουργία της Όλαφ και το θέμα του ΙΠΠΟ, του θα το δούμε σε επόμενη φάση. Πάντως συνεργαζόμαστε στενά με, την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ και στο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν για το ΙΠΠΟ προβλέπονται το 12 ορισμένες δραστηριότητες και το 13. Τώρα γίνονται μόνο προκαταρκτικές συζητήσεις για, το, για τον ρόλο του ΙΠΠΟ και τις σχέσεις μεταξύ ΙΠΠΟ και Όλαφ. Μάλλον είναι πρόωρο ακόμη να καθορίσουμε πλήρως από τώρα ποιο ακριβώς θα είναι η σχέση μεταξύ Όλαφ και ΙΠΠΟ. Ούτως ή άλλως όμως το θέμα θα ξανασυζητηθεί εδώ στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο διότι το ΙΠΠΟ είναι πολύ λεπτό θέμα και πρέπει μαζί να τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριος Πατρικιαήλη. Πρόεδρε, Ήθελα να εμβαθύνουμε στα θέματα αυτά, αλλά θα περιμένω την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ζητήσατε το λόγο, η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει την άποψή του για πάρα πολλά θέματα ήδη από τον Νοέμβριο του 2008. Πρώτη ανάγνωση. Σε, δύο, σε λίγο θα κλείσει διετία, θα έχει τα γενέθλιά της η πρώτη ανάγνωση. Και πέρσι είχαμε τη δεκα... δεκάτη επέτειο της Όλαφ. Και εγώ έβαλα στοίχημα ότι μέχρι τα 20 χρόνια δεν θα είχε λύσει το θέμα ε, της ε, νομικής βάσης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να το παραπέμψουμε στις καλένδες. Εντάξει, να συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα, αλλά εμείς την άποψή μας την έχουμε καταθέσει. Τι να συμμετέχουμε, να ξαναπούμε τη γνώμη μας σε δεύτερο γύρο. Εντάξει, μπορεί να αλλάξουν λεπτομέρειε, αλλά επί τη ουσία η θέση του Κοινοβουλίου είναι δεδομένη. Μπορούμε να κρατήσουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ, γιατί έχουμε και επιχειρήματα που τα στοιχειοθετούν αυτά. Δεν θα πω ότι η είναι στο Συμβούλιο ε, και θα πρέπει να μεταφερθεί στο Κοινοβούλιο. Γιατί επειδή οι μεν δεν ξέρουν τι θέλουν να τσακωθούν και οι δε, όχι, εμείς τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε βάλει κάτω και για όσους αναγνώστες ενδιαφέρονται έχουμε 11 έγγραφα εργασίας παρακαλώ, 11 και ε, στην ιστοσελίδα της Κοκομπίου από την περασμένη θητεία και είμαι πρόθυμα να το στείλω σε όποιον ενδιαφέρεται. Τώρα δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση αέναη για τη μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης. Επειδή είναι απρόθυμο το Συμβούλιο και θέλει να χρονοτριβεί, να κολυσιεργεί και να διονύζει τη συζήτηση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την εμπλοκή του Συμβουλίου. Δεν θα την ξεπεράσουμε με το ξαναρχίσουμε εμείς ολόκληρη συζήτηση επάπειρο. Το Κοινοβούλιο έχει άποψη. Λοιπόν, παρακαλώ να πάρετε τα πράγματα στα χέρια σας, στοχευμένα, με νομοθετικό πρόγραμμα. Έχετε κάνει πρόταση, εμείς την τροποποιήσαμε. Τώρα θέλετε να κάνετε νέα πρόταση και να ξανααποφανθούμε. Θα χάσουμε άλλα δύο χρόνια περίπου και ακόμα δεν θα έχουμε κερδίσει τίποτα σε ουσία για τη μεταρρύθμιση και μάλλον το Συμβούλιο θα είναι ακόμα απρόθυμο. Η πρόταση λοιπόν υπάρχει νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάνω σε αυτή δεν μπορούμε να μπούμε στη διαβούλευση με το Συμβούλιο και να αγαθήσουμε να τα βάλουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε. Και έχουμε και προτεραιότητες και άλλα πράγματα που δεν είναι του παρόντος. Α μην τι άλλο να αρίσουμε το γενικό διευθυντή, να του δώσουμε ένα πληρωτή. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα στην νομική βάση. Δεν θέλω τώρα να φέρετε νομοθετική πρόταση νέα, γιατί αυτό θα χρειαστείτε πάρα πολύ χρόνο. Και εσείς και εμείς. Και μέχρι τα τέλη του έτους αυτό αποκλείεται. Λοιπόν, να το πω και αυτό από την αρχή. Άλλωστε, ο στόχος της συζήτησης ανακαθέν αυτός ήταν. Στο σημερινό νομοθετικό κείμενο να βασιστούμε και να αρχίσουμε τις διαβουλεύσεις. Αυτό είναι το ένα που θέλω να ξεκαθαρίσω. Ένα δεύτερον. Έχω θορυβηθεί από αυτά που μας είπατε για την επιλογή του Γενικού Διευθυντού. Στη νομική βάση λέγει concertation. Concertation, όχι consultation. Δεν είναι απλή έτσι, πρόταση. Είναι συνεννόηση. Δεν ξέρω αυτή η μετάφραση αγγλική. Σε όλες τις άλλες γλώσσες λέει concertation. Και η αρχική τότε εκδοχή πριν από 10 χρόνια ήταν τα γερμανικά. Και έλεγε συνεννόηση και όχι απλή διαβούλευση, έτσι μια συζήτηση κοινή και να γίνει αυτή η συνεννόηση. Concertation. Την περασμένη φορά είχαμε 5-6 υποψηφίους, τους ακούσαμε και απεφάνθημε. Δεν θέλω τώρα να μας φέρετε 2-3 και να μας πείτε ωραία διαλέξτε. Όχι να μην αποκλίνουμε από την περασμένη διαδικασία και δεν υπάρχει και λόγος κατά την άποψή μου να αλλάξουμε τώρα μέθοδο. Αυτή θα ήταν η δεύτερη παράκλησή μου και έρχομαι τώρα στην τρίτη παράκληση. Ε, την ε, εισαγγελία, το EPPO το περίφημο, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι θα το κάνουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ ανησυχώ βαθύτατα. Αν περιμένουμε να έρθει ο Ευρωπαίος εισαγγελέα, θα ξεχάσουμε το 5 και στο χέρι και θα είμαστε στο 10 και καρτέρι. Περίμενε, μπορεί να φτιάξουμε και εισαγγελέα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει αυτή η βαριά, άκαμπτη, σούπερ δομή, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας ποντάρει στη Eurojust για τον εισαγγελέα και όχι ε, στην Όλαφ. Η Όλαφ είναι ο μέγας χαμένος ε, της συνθήκης Λισαβόνας και αν έρθει τώρα μια νέα ευρωπαϊκή δομή που θα αποτύχει, θα έχουμε δύο αποτυχημένες ε, δομές παρά να έχουμε φτιάξει τη μία που έχουμε τώρα και να λειτουργήσει. Δεν είναι ότι αγαπάω πολύ την Όλαφ, αλλά μετά από 10 χρόνια επιτέλους είναι θεμητό να έχουμε την αξίωση να λειτουργεί σωστά ένα πράγμα που φτιάξαμε πριν από 10 χρόνια. Και το θέμα δεν είναι να βάλουμε το πρόβλημα και να πούμε καλά κάποια ώρα θα έρθει και ο εισαγγελέα και θα λυθεί, σιγά μη Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Σας ευχαριστώ να προσθέσω και εγώ μια δική μου παρατήρηση. Μου φαίνεται ότι διαφαίνεται η πολιτική βούληση όλων των ομάδων εδώ, της Επιτροπής μας Ελέγχου του Προπολογισμού, όχι μόνο να διατηρήσουμε μια όλα, με κύρος και θεσμικός με ένα ρόλο σημαντικό, αλλά επιπλέον η ικανότητα δράσης της να ενισχυθεί. Το επιβεβαίωσαν και οι δύο σημαντικές επισκέψεις που κάναμε στην Ελλάδα και την Κροατία. Και παληθεύσαμε και σε άλλα κράτη της Ένωσης και το έδειξε αυτό η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας ότι υπάρχουν εδώ προβλήματα. Η Όλαφ λοιπόν μπορεί να καταπολεμήσει την απάτη που υπάρχει στις χώρες. Το οικονομικό συμφέρον των πολιτών της Ένωσης σημαίνει όχι μόνο καταπολέμηση της απάτης, αλλά και καταπολέμηση των, ε, της παρανομίας και να βεβαιωθούμε ότι αυτό που σημαίνει τα τελευταία χρόνια, η κερδοσκοπία δηλαδή, που έχει βρει στα δημόσια κρατικά κονδύλια έναν τρόπο να πλουτίσει, να εμποδιστεί. Και πολλές φορές αυτό έχει διαπεράσει και στα θεσμικά όργανα, διότι η διαχείριση των δημοσίων κονδυλίων πολλές φορές έχει να κάνει και με τους θεσμούς, με, το, με τις αρχές. Έτσι λοιπόν πλήττεται ο ιστός, ο δημοκρατικός ιστός των ε, χωρών. Σε αυτή λοιπόν τη φάση νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την Όλαφ, γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε και να δούμε, ώστε να φροντίσουμε η συζήτηση για το Γενικό Εισαγγελέα και για τη Eurojust να μην ε, αφήσει στο παρασκήνιο την ε, όλα. Αυτό έχω πει αυτό και σε κάποιες άτυπες συνομιλίες με συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Έχω την εντύπωση ότι κάποιες προσ... Ε, κάποιοι προσπαθούν να περιοριοποιήσουν τον ρόλο της Όλαφ με αφορμή τον, τη Γενική Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που είναι σημαντικό στόχος, πρέπει να το επιδιώξουμε Όμω σήμερα συζητούμε για την Όλαφ που ήδη είναι ένα πιο προχωρημένο σχέδιο σε σχέση με τον Γενικό Εισαγγελέα. Έπειτα, ακούμε τι επιτροπέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω βουλευτέ, βεβαίω θα φροντίσουμε να έχουμε και τι κατάλληλε κοινοβουλευτικέ απαντήσει, ώστε να εναρμονιστεί ο ρόλο των θεσμικών αυτών οργάνων. Νομίζω σε κάθε περίπτωση οι πολίτε αυτό που μα ζητούν είναι διαφάνεια. Διαφάνεια και για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τη διαχείρισή του διότι υπάρχει όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ως προς τη διαχείριση των κονδυλίων τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για δις ευρώ και δημόσια κονδύλια. Έτσι λοιπόν, Επίτροπε, ίσως σήμερα να μπορούσατε να μας δώσετε μια πιο συγκεκριμένη συνεισφορά Και εμείς από τη δική μας Επιτροπή θα φροντίσουμε τη φωνή μας να την υψώσουμε ώστε η Όλαφ να παραμείνει ανεξάρτητη και με κύρος και ελπίζουμε οι αρχές αυτές που και εσεί εκφράσατε να μεταφραστούν σε συγκεκριμένε δράσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Σεμετά. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, για το έγγραφο αυτό και για την τήρηση, την υποδειγματική τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των υποσχέσεων που είχατε δώσει εδώ στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων για το έγγραφο το ίδιο για την επιλογή του Γενικού Διευθυντού τώρα, σε σχέση με τα όσα μας είπατε, θα προσπαθήσω να τα φέρω αυτά κοντά στο κείμενο. Είπατε, στις 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε υποψήφιο και μετά είπατε shortlist, ένα σύντομος κατάλογος, τουλάχιστον εγώ αυτό άκουσα από τη γερμανική καμπίνα. Στις 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν τι θα έχουμε, ένα μοναδικό υποψήφιο, μήπως κάνατε λάθος ε, και δεν νοούσατε αυτό γιατί εγώ θα περίμενα να έχουμε μια σειρά υποψηφίων ε, ενδεδειγμένων ε, που θα μας απασχολούσαν ενδεχομένως. Η Επιτροπή μας έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει το έχουμε συζητήσει και στο θέμα του προσωρινού διευθυντή, αυτό που είπε η κυρία Γκρέλσλε, αν είναι consultation ή concertation, εκεί να δείτε ώρες που έχουμε αφιερώσει οι συντονιστές σε αυτό το θέμα. Και είναι σαφής νομίζω η κατάσταση και το συμπέρασμά μας. Δεν μας ακούτε απλώ τη γνώμη μας, δεν είναι διαβούλευση, ε, ε, έχουμε λόγο. Και θέλουμε να ασκήσουμε τη δυνατότητα αυτή που έχουμε, γιατί όσο λιγότερους υποψηφίους μας φαίνεται, τόσο λιγότερο λόγο θα έχουμε. Να το πω ηρωνικά. Η επιλογή όταν έχουμε δύο είναι διαφορετική από όταν έχεις, ξέρω εγώ, τέσσερις-πέντε, για να πω ένα νούμερο έτσι. Εξ όσων γνωρίζω έχει προχωρήσει σχετικά η διαδικασία και την προπερασμένη εβδομάδα έγιναν και συνεντεύξεις με 11 υποψηφίους παρακαλώ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνει η υπόθεση και κοντά στο κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι, όπου θα έχουμε ένα επαρκή αριθμό υποψηφίων για να μας παρουσιάσετε και στο κοινοβούλιο. Θα το θεωρούσα πολύ σημαντικό και παρακαλώ να το σχολιάσετε. Θα θεωρούσα, λέω, πολύ σημαντικό τους υποψηφίους, άνδρες και γυναίκες, να τους έχουμε και εμείς υπόψη μας και να έχουμε την ευκαιρία να τους ε, ακούσουμε εκτενώς, να λάβουν θέση, να μας πούν τι σκέφτονται ε, για τη θέση του Κοινοβουλίου που υπάρχει και είναι γνωστή και τι άλλες προτάσεις, ιδέες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν στο έγγραφο προβληματισμού σας. Νομίζω θα ήταν αυτή μια πολύ καλή συζήτηση και καρποφόρα και κάνει τη διαδικασία και διαφανή, αλλά θα έχουμε και σαφή αντίληψη για το τι μέλη γενέστε και τι πορεία παίρνει η Όλαφ. Και θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε και τη δημιουργικότητα, ας πούμε, των υποψηφίων. Με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Grazie να δώσουμε τώρα το λόγο στον ε, Επίτροπο Σεμέτα, αν θέλει να απαντήσει. Thank ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω με το τελευταίο ερώτημα. Για να αποσαφινιστούν τα πράγματα. Μάλιστα, θα λάβετε κατάλογο υποψηφίων και θα μπορέσετε να θέσετε ερωτήματα σε όλους τους υποψήφιους του καταλόγου για την τελική τους έγκριση και διορισμό. Αυτό δεν είναι, πρόβλημα. Σε αυτή τη φάση Κοιτάζουμε ακόμη τα τυπικά δηλαδή, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για να δούμε ποιους θα βάλουμε στον κατάλογο. Οι υποψήφοι που θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από το CCN ή μέσω του CCN θα γίνουν δεκτοί για εξέταση και θα δούμε μετά αν θα γίνουν δεκτοί και ως υποψήφοι για να υπάρξει ο τελικός κατάλογος υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντού. Και τότε θα αρχίσει και η συμβολή του Κοινοβουλίου και του Συμβολίου στην διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντού. Νομίζω ότι δεν έχουμε διαφορά απόψεων εδώ. Συμφωνώ να είναι τελείως διαφανής η διαδικασία ώστε να είναι βέβαιο ότι θα επιλεγεί ο καλύτερος ως Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Γιατί και αυτό είναι κοινό μας συμφέρον. Να έχουμε μια Όλαφ δηλαδή που να λειτουργεί όπως πρέπει. Τώρα οι άλλες ανησυχίες της κυρίας Γκρέσλερ για τα διαδικαστικά, για τη συνέχεια, θα ήθελα να της πω ότι δεν υπονοούσα τη νέα διατύπωση της πρότασης της Κομισιόν απλώς, απλώς με βάση αυτά που είπατε, τις αντιδράσεις σας στο έγγραφό μας, ήθελα απλώς να ενημερωθεί η πρόταση της Κομισιόν, που είναι από το 2006, να εξυγχρονιστεί και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν είμαστε αποτελεσματικοί, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε με την ενημερωμένη πρόταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Και έτσι να τελειώσει όλη η διαδικασία το επόμενο έτος. Επίσης εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος ως προς την κατάσταση που επικρατεί στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι το Συμβούλιο προτίθεται να συνεδριάσει η ομάδα εργασίας του δηλαδή στις 28 Σεπτεμβρίου για να συζητήσει το εγγραφό μας και θα κάνω όλες τις προσπάθειες που χρειάζονται για να διασφαλιστεί ότι και στο Συμβούλιο θα πάνε τα πράγματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να έχουμε και τις δικές τους απόψεις όσο το δυνατόν συντομότερα. Τώρα για το ΙΠΠΟ. ΙΠΠΟ για τον Ισαγγελέα. για τον Ισαγγελέα που λένε. Είχα πει ότι πρέπει τώρα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην Όλαφ και να τελειώσουμε τη μεταρρύθμιση της όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ότι αποκλείουμε και κάποια προπαρασκευαστική δουλειά για την εισαγγελία ΠΠΟ. Διότι χρειαστεί χρόνος, χρειάζεται πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή συζήτηση, συμφωνία μεταξύ κρατών, μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων. Πρέπει να γίνει κάποια προπαρασκευή και για εκεί. Αλλά τώρα επικεντρωνόμαστε στην Όλαφ κυρίως. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να καταλήξει η διαδικασία. Όσο δυνατόν συντομότερα όπως ξαναείπα και για τις δικές σας ανησυχίες κύριε Πρόεδρε να συμφωνώ ότι το θέμα της δωροδοκίας και διαφθοράς είναι επίσης σημαντικό, όλα είναι σημαντικά. Και πρέπει και αυτό να εμφαίνεται και να εμφανίζεται στον κανονισμό της Όλαφ. Επαναλαμβάνω διαφθορά δωροδοκία. Όπως και με τις απάντες, όπως με τις απάτες να ασχολείται και με τη δωροδοκία. Να, σύντομα αυτά είχα να σας α, συνοψίσω και, και ελπίζω η αντίδρασή σας στο έγγραφό μας να είναι σύντομη και να αν χρειαστεί, αν χρειαστεί να ξαναέρθω να τα πούμε είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας άμα θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες να περιγράψω του εγγράφου γιατί έχει πολλές σημαντικές λεπτομέρειες το παραδέχομαι και ίσως χρειαστεί και άλλη ανταλλαγή απόψεων και για τις λεπτομέρειες αυτές εγώ μπορώ να ξανάρθω δεν με πειράζει αυτό Ευχαριστούμε και εμείς από την πλευρά μας. Είμαστε διαθέσιμοι ώστε να περάσουμε στη συζήτηση και για τις επιμέρους προτάσεις τροπολογίας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν Επίτροπε και σας αποχαιρετούμε και περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Απαλλαγή 2008, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Το λόγο έχει η κυρία Ματιέ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε γιατί αποφασίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις 7 Μαΐου 2010 να αναβληθεί η απόφαση απαλλαγής του 2008 για την Αστυνομική Ακαδημία. Τώρα, συνάδελφοι, θα δούμε τι πρόοδος επιτέλεσε η Ακαδημία αυτή για να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και δημοσιονομική της διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο το Κοινοβούλιο έχει απευθύνει πολλά αιτήματα προς την ε, Ακαδημία και εγκρίθηκε και απόφαση με την απόφαση του 2008 στην Ολομέλεια. Έτσι, λάβαμε από το διευθυντή της ΕΠΟΛ, της Αστυνομικής Ακαδημίας, ε, διευθυντής που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του από τις 16 Φεβρουαρίου 2010, ένα διοικητικό πολιετές πρόγραμμα για το 2010-2014 και μια έκθεση υλοποίηση των δράσεων των προβλεπόμενων επιχειρήσεων για το 2010. Θα ήθελα να στραφώ στη θέση του διευθυντού αυτής της Ακαδημίας, τον κύριο Μπάνφη, αν νομίζω ότι έχει φτάσει και στην αίθουσα, Κύριε Διευθυντά, στην απόφαση που συνοδεύει την απόφαση αναβολή τη ε, απαλλαγή τη Ακαδημία, εδώ ενημερώνουμε τι αρχέ απαλλαγή για τα αποτελέσματα των ερευνών που έγιναν στην ε, Όλαφ. Ε, και θα θέλαμε να ξέρουμε επίση γιατί ε, ήταν αυτά τα πορίσματα τη έρευνα. Επίση, σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΠΟΛ, τη Αστυνομική Ακαδημία και μετά την έρευνα τη Όλαφ, καμία διοικητική ποινή δεν ε, επευλήθη στους, ε, σε όσου είχαν υποπέσει σε παραπτώματα. Θα θέλαμε να μα ενημερώσετε και σε σχέση με το θέμα αυτό. Και σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των δημοσιονομικών πρακτικών τη Ακαδημία. Αναφέρεται στην ενημερωτική επιστολή τη Αστυνομική Ακαδημία για το 2010 ότι ε, οι εσωτερικέ. Ότι στις 12 Μαΐου 2010 οι εσωτερικές ε, υπηρεσίες ελέγχου της Επιτροπής πρότειναν την οργάνωση σεμιναρίων για την βελτίωση των ε, αρμοδιοτήτων της ΣΕΠΟΛ για την για, τον, για την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτή η κατεπίγουσα μερίδα εκπαίδευσης έλαβε χώρα. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα θέλαμε να ξέρουμε αν έχει καταφέρει, μάλλον αν καταφέρατε να λάβετε υπόψη το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί για τον Ιούλιο του 2010 και θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει έρευνα από εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές ε, για τον προβλογισμό σα του 2009. Θα σας αφήσω για την ώρα να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα και μετά θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Τώρα το την λόγο έχει διευθυντή της αστυνομική Ακαδημίας. Dear Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφραστώ εδώ ενώπιόν σας και να σας χορηγήσω την ενημέρωση αυτή και τις απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Κυρίες μου και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς σύντομα να κάνω μια εισήγηση μάθατε ότι ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 16 Φεβρουαρίου. Προηγουμένως είχα περάσει 30 χρόνια σε αστυνομικές δουλειές στην Ουγγαρία. Άρχισα από το δρόμο και κατέληξα ως αντιδιευθυντής ή υποδιευθυντής της αστυνομίας. Τα τελευταία χρόνια Ήμουν υπεύθυνο για την επιτήρηση των συνόρων και άλλα διεθνή και διαμεθοριακά θέματα. Στη νέα μου θέση άρχισα πρώτα να μελετώ πώς είχαν τα πράγματα, γιατί δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Χρειάστηκε νέα διαχείριση της κρίσης, ιδιαίτερα της καλής διαχείρισης της υπηρεσίας. Ως προς τα συγκεκριμένα σας ερωτήματα απαντώ τα εξής. Η έρευνα της Όλαφ δεν είναι δημόσια και άρα τα αποτελέσματά της δεν δόθηκαν στον διευθυντή της Ευρωάστα και η συζήτηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων της έγινε αποκλειστικά μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν δικαίωμα ψήφου. Οι απόρριτες αυτές έρευνες, οι απόρριτες έρευνες για τον Διευθυντή του ΣΥΠΟΛ δεν προβλέπουν απαντήσεις να δοθούν. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχω πνεύμα συνεργασίας μεταξύ σας. Προς δεν μου επιτρέπετε. Όσα τη δημοσιονομική διαχείριση τη διήμερη εκπαίδευση του προσωπικού δηλαδή, αυτό εφαρμόζεται σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση 16 με 17 Ιουνίου με συμμετοχή του Διευθυντή του Δημοσιονομικής Μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών από την Κομισιόν και τη διεύθυνση της ΥΠΟΛ και τη δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί αυτή την εβδομάδα 15 και 16 Ιουνίου λέει ο μιλητής. Ιουλίου δηλαδή. Αυτή η διφασική εκδήλωση λοιπόν θα συμπεριλαμβάνει τον προγραμματισμό και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και εκμάθηση των βελτίστων πρακτικών στην Ένωση. Την πρώτη ημέρα της μετεκπαίδευσης αυτής ή της ημερίδος ή του σχεδιασμού γιατί είναι και τα δύο, ο πρόσωπος της Κομισιόν της Υπηρεσία Εσωτερικού Δημοσιονομικού Ελέγχου και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν προσκληθεί. Και ο διευθυντής της ΥΠΟΛ θα εξηγήσει τον νέο σχεδιασμό. Και τη δεύτερη ημέρα θα συνεχίσουν τα ίδια αλλά με ειδικευμένε ομάδες και εργαστήρια για να δούμε πιο συγκεκριμένα τι προγραμματισμός χρειάζεται για το 12 και εν μέρη και για το 11. Πρώτα το 11 μετά το 12. Όσο για τις εκθέσεις των εισηγητών θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτές, θα υπάρχει. Το 2009, οι προϋπολογισμοί του 2009 για τη ΣΥΠΟΛ έγιναν δεκτοί από το, δημοσιονομ... από το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο είχε ήδη δηλώσει ότι στην ιστορία της Ήπολ για πρώτη φορά μπόρεσε να μας δώσει λογαριασμούς που να συμφωνούν με το δημοσιονομικό κανονισμό. Τώρα τι θέλετε να συνεχίσω έτσι με τη σύντομη σύνοψη ή μόνο με τις απαντήσεις των ερωτήσεων. Αυτό θέλω να μου πείτε. Αυτό. Θα μπορούσατε να μου πείτε περισσότερα για την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο της απόφασης για το 2009. The European Court of Auditors το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έκανα την έρευνα του πρώτου τομέα στην Αστυνομική Ακαδημία μεταξύ επιτόπια έρευνα μεταξύ 1η και 8 η Μαρτίου 2010 για τις δράσεις της ΣΕΠΟΛ και τα πρώτα πορίσματα ήταν ότι υπάρχουν μεγάλα σφάλματα στους λογαριασμούς της Αστυνομικής Ακαδημίας που δεν είναι αποδεκτή σε αυτή τη φάση. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια εντατική προσπάθεια για τους προσωρινούς μας λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου το διορισμό συμβούλων από την πλευρά των δημοσιονομικών θεμάτων και με την στήριξη των ανθρωπίνων πόρων μας για να ε, δούμε γιατί υπήρχαν αυτά τα σφάλματα και οι ελλείψεις που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο. Μετά από αυτή την εντατική, όπως είπα, προσπάθεια, υποβάλαμε τη διορθωμένη εκδοχή στο ελεγκτικό συνέδριο. Τότε έγινε ένας δεύτερος έλεγχος στο Μπρέμσχιλ μεταξύ 28 Ιουνίου και Δευτέρα Ιουλίου και τα πορίσματα της έρευνας αυτής ήταν ότι πλέον οι λογαριασμοί μας ήταν οι Κύριε Δευθυντά, το 2008 αστυνομική η Ακαδημία έπρεπε να μεταφέρει 2,30 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2% του συνολικού της προπολογισμού. Τι μέτρα προβλέπονται εδώ, γιατί το κολέγιο προτείνει τα κονδύλια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο τέλο της χρονιάς να χρησιμοποιηθούν ω αποθεματικό για επόμενη χρονιά. Αυτή η στατηγική, κατά την άποψή σας είναι η καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκε της σημερινέ και με βάση το την απόφαση της, ε, της αρχής της εξειδίκευσης. Οι πιστώσει επίση σωστά χρησιμοποιήθηκαν ε, για τι προβλεπόμενε δράσει και η συμμετοχή των κρατών μελών στι δράσει τη Αστυνομική Ακαδημία δεν έχουν μειωθεί τα τρία τελευταία χρόνια. Τι μέτρα έχετε σχεδιάσει μετά από αυτέ τι διαπιστώσει, και πιστεύετε ότι από αυτέ τι προποθέσει μπορεί να διευρυνθεί η εντολή και αποστολή τη ε, Όλαφ. Εδώ της ΣΕΠΟΛ εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κατάλογος των μελών της ΕΠΟΛ ε, με, τη, με τα στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και επίσης πρέπει να φαίνεται ποιες δράσεις θα προβλέψει η Ακαδημία. Μπορείτε να μου πείτε γιατί υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις ή να μου πείτε αν σκοπεύετε να γίνει κάτι γι' αυτό σύντομα. Καταρχάς, θα πρέπει ειλικρινά να πούμε ότι ο δημοσιονομικός σχεδιασμός του ΣΥΠΟΛ ε, της ε, Αστυνομικής Ακαδημίας ήταν εσφαλμένος. Δηλαδή, διαφορετικές δραστηριότητες ε, είχαν υπερβολική πρικοδότηση και τελικά πολύ χαμηλή απορρόφηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το 2008 χαρακτηρίζει την κατάσταση από την αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Και δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι αυτή η υποπορρόφηση δεν πρόκειται να λήξει τελείως μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ελπίζω να κάνουμε πρόοδους και λογικές. Σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες και κανονισμό, τα ποσά που δεν απορροφήθηκαν φέτος αλλά είναι ε, δεσμευμένα, μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος και μπορούν να ε, δαπανηθούν αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο είχαν εγγραφεί και όχι μεταφορές πιστώσεων για άλλους σκοπούς. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η ΣΥΠΟΛ δεν ήταν σε θέση να κάνει αναδιάταξη των πόρων από το 2008 στο 2009 και η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια από το 2009 την προσμεταφορά το 2010. Θα πρέπει ε, τα χρήματα ε, να ε, πιστωθούν εκεί που έχουν αναλυφθεί υποχρεώσεις. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Ακαδημία θα πρέπει να βελτιώσει τη διοικητική της λειτουργία και δυνατότητα αναθεωρώντας την παρούσα δομή με ε, οργανωτικές αλλαγές ε, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο στις 25 Μαΐου αποφάσισε νέα οργανωτική δομή και διάρθρωση, που ακολουθεί τις συμβουλές ή συστάσεις των ελεκτών, συμπραβανωμένης και της εσωτερικής υπηρεσίας οικονομικού ελέγχου, αλλά και του ελεγκτικού συνεδρίου. Δηλαδή, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε ε, τη γραμματεία ως προς τα οικονομικά της ένα μέρος. Είναι μικρή μονάδα και σύμφωνα με το μέγεθος ε, της δομής είναι υπερβολικά αποκεντρωμένη η οικονομική διαχείριση. Λοιπόν, από την πρώτη πρώτου θα έχουμε οικονομική μονάδα που κεντρικά θα διαχειρίζεται το προπολογισμό και θα ελέγχει, θα παρακολουθεί σωστά, θα έχει υποπτία ε, των πιστώσεων και πού διατίθενται, το σύνολο του προπολογισμού εννοώ και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και το νομικό εργαλείο που λέγεται μεταφορά πιστώσεων για να ε, απορροφηθούν τα κονδύλια καλύτερα. Άλλο τώρα θέμα. Για το έτος 2010, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, ε, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του παρελθόντος, ιστορικές αναφορές, ας πούμε, για να ε, απορροφώνουν καλύτερα τα κονδύλια. Σε αυτό φορά τώρα τη συμμετοχή της μετακπαίδευσης και της, ε, της ε, κατάρτισης, αναλύουμε το πώς συμμετέχουν τα διάφορα κράτη-μέλη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ακαδημίας. Είναι γεγονός ότι φθήνει η συμμετοχή των κρατών μελών για τους εξής λόγους. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη ενημέρωση εξυγχρονισμού των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών και το αντικείμενο της αστυνομικής ακαδημίας. Υπάρχουν μερικέ αλλαγέ όπως είναι η συνθήκη τη Λισαβόνα, το πρόγραμμα τη Στοχόλμη και το πρόγραμμα δράση η ε, ολοκληρωμένη στρατηγική ασφαλείας. Όλα αυτά είναι θέματα που στρέφουν σε μια νέα κατεύθυνση την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Δηλαδή, θα αρχίσει τις επόμενες ημέρες ένας νέος προγραμματισμός και το 2011 θα πρέπει η Αστυνομική Ακαδημία να εμφανίσει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι διάφορες επιμέρους αποφάσεις που συζητώνται σε διάφορε ομάδε εργασία και άλλε επιτροπέ. Όλα αυτά τα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μα. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο ή τα ονόματα του Διοικητικού Συμβουλίου, το συζήτησε και αποφάσισαν ότι δεν δημοσιεύουν τα ονόματα των μεμονωμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι όλα τα υπόλοιπα όργανα, οι υπόλοιποι οργανισμοί σε αυτό το κλάδο, η Europol, η Frontex, δεν ε, δημοσιοποιούν κατάλογο μελών των διοικητικών συμβουλίων. Πέρα από αυτό όμως, είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει καλή ενημέρωση και διαφάνεια και νομίζω αυτή διασφαλίζεται από τα όσα δημοσιεύονται στην ισοσελίδα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άλλοι συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Αν όχι, παρακαλώ. Η κυρία Κρέσλε. Θα ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Όλαφ, να δούμε τι κάνει. Και το ελεκτικό συνέδριο θα ήταν καλό να ακούσουμε για να μάθουμε τι έγινε το 2009. Ίσως και τον εσωτερικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλούμε, εκπρόσωπος της Όλαφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Γκρέσλε, η Όλαφ, όπως γνωρίζετε, υπέβαλε έκθεση με έναν αριθμό πορισμάτων σε σχέση με τις ατασταλίες που διαπιστώθηκαν στο φάκελο της Αστυνομικής Ακαδημίας που αφορούσαν αρκετά άτομα αλλά και την υλοποίηση οικονομικών και δημοσιονομικών δομών. Η έρευνα αυτή περατώθηκε με ένα κεφάλαιο πειθαρχικό, το οποίο ο νέος διευθυντής σας εξήγησε ότι τελικά δεν οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων και το φάκελο αυτό τον αποστήλαμε και στις δικαστικές αρχές της Βρετανίας που αυτή τη στιγμή ακόμη εξετάζουν το όλο θέμα, την υπόθεση. Έτσι λοιπόν η υπόθεση αυτή ακόμη εκδικάζεται από τις Βατανικές Αρχές, οπότε δεν είμαστε και σε θέση να δώσουμε περιττέρω πληροφορίες. Υπήρχε βεβαίως και το κεφάλαιο της ανάκτησης, των ανακτήσεων, το οικονομικό κεφάλαιο και ως προς αυτό ζητήσαμε να υπάρξει προσεκτική εποπτεία προσεκτική παρακολούθηση και καταγράφω εδώ προσεκτικά όσα ακούσαμε γιατί φαίνεται να υπάρχει πρόοδος, τόσο το καλύτερο. Ελπίζω ότι θα ανακτήσουμε το σύνολο των ποσών μας λείπουν και έτσι θα αρχίσουν να λειτουργούν σωστά οι δομές. Σημείωσα όσα είπε ο νέος διευθυντής περί της κατάστασης που κληρονόμησε η οποία δεν ήταν ε, και τελείως ε, καταπληκτική. Αυτό όντως επιβεβαιώνει και τα δικά μας τα πορίσματα. Έπρεπε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Και εδώ μιλάμε κυρίως για την διόρθωση των ε, δημοσιονομικών λογαριασμών ως προς την έκθεση της Όλαφ. Απεστάλλει στο Governing Board, στο Διοικητικό Συμβούλιο, και απευθύνθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα. Η Όλαφ είναι ένας ελεγκτικός οργανισμός περιορισμένος που πρέπει να δράσει μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι φέραμε εις πέρα στα καθήκοντά μας και καταγράφουμε με ικανοποίηση τις εξελίξεις που μας ε, ανακοινώθηκαν σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Γκρέφλε. Ζητώ συγγνώμη που θέλω να ρωτήσω ξανά τον εκπρόσωπο της Όλαφ. Ε, μήπως κατάλαβα μόνο τα μισά από αυτά που είπατε. Λέτε ότι δεν, θα, δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Δηλαδή, ποιος θα τις επέβαλε, το Διοικητικό Συμβούλιο υποθέτω. Σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο διευθυντή, τι απέγινε. Γιατί. Νομίζω ότι όλα διαλύονται σε μια συγκεχημένη αδράνεια. Και ποια είναι, δεν υπάρχει θέμα πειθαρχικού εδώ, πραγματικά το έχει ξεχάσει ο κανονισμός, θα πρέπει να διορθωθεί στον επόμενο ε, κανονισμό. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιο να επιβάλλει και κυρώσεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Ποιε από τι συστάσει τη Όλαφ ε, έχουν εφαρμοστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ποιε όχι και αν όχι γιατί. Αλλά παρακαλώ πρώτα να μα απαντήσει ο εκπρόσωπο τη Όλαφ. Παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Σημειώνω τις ερωτήσεις σας κυρία Γκρέσλε. Όμως η Όλαφ δεν μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα είναι, οφείλει να κάνει. Δηλαδή να εξαγάγει μια έρευνα. Είναι διοικητικό θέμα αυτό, διοικητική έρευνα διατυπώνει κάποιες συστάσεις στη συνέχεια και δεν είναι δική της αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Ε, θα γνωρίζετε ότι είμαστε ένα θεσμικό όργανο που δεν έχει τέτοιου είδους εξουσίες. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και όντως το πράξαμε είναι ότι ενημερώσαμε τις αρχές τι ενδιαφερόμενε αρχέ ότι θα έπρεπε εκείνε, εφόσον το ήθελαν, να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, να επιβάλλουν τι ενδεχόμενε κυρώσει. Σε ό,τι αφορά το νομικό, το δικαστικό θέμα, το εξετάζουν αυτή τη στιγμή οι αρχές της Βρετανίας και εκείνες εφόσον το κρίνουν λογικό θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Σε ό,τι αφορά το πειθαρχικό σκέλος. Είναι ενδιαφέρον το ζήτημα, διότι για άλλη μια φορά τίθεται το πρόβλημα το πειθαρχικό σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Λόγου χάρη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει ένα πειθαρχικό ζήτημα, είναι πολύ απλό να παραπεμφθεί στην ΙΝΤΟΚ, η οποία θα ασχοληθεί με την πειθαρχική διαδικασία. Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλα τα θεσμικά όργανα. Κάποιες φορές το να δημιουργηθεί πειθαρχικό συμβούλιο προκαλεί για τρεις δυσκολίες σε άλλα θεσμικά όργανα. Διοικητικές δυσκολίες, τεχνικές, γιατί χρειάζεται στο, η συμμετοχή στο συμβούλιο, αυτό μελών που πρέπει να έχουν βαθμό από 15 κάποιες φορές έως και 16 και δεν το έχουν αυτό όλα τα μέλη αναγκαστικά. Οπότε είναι θέμα η δημιουργία πειθαρχικών συμβουλίων στο επίπεδο των οργανισμών. Εδώ θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα διοργανικό ενδεχομένω πειθαρχικό συμβούλιο που να εξυπηρετεί όλου. Αλλά το πρόβλημα είναι οξύ και δεν είναι αυτή η οριστική λύση και δεν την έχουμε ακόμη αποφασίσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση της Αστυνομικής Ακαδημίας, κάναμε το μόνο που μπορούσαμε, δηλαδή να αποστείλουμε, να παραπέμψουμε το ζήτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει ή όχι πειθαρχικέ ποινές ή κυρώσεις, όπως κάνει ένα πειθαρχικό συμβούλιο. Μόλις μας το είπε ο νέος διευθυντής όμως, καμία κύρωση δεν επιβλήθηκε στους ενδιαφερομένους. Αυτό δεν μπορώ παρά να το καταγράφω από την πλευρά της Όλαφ. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, όπως σας είπα, να επιβάλλουμε κυρώσεις. Μπορούμε να τις συστήσουμε. Να συστήσουμε την παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο ή την ε, οικονομική ανάκτηση, αλλά δεν είμαστε εμείς ποτέ ε, ο υπεύθυνο για την επιβολή των κυρώσεων. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνω... Να στήσω το δύο Να δούμε την έκθεση, να τη διαβάσουμε ε, στο δωμάτιο ασφαλείας που είναι και κλεισμένο των θυρών και να δεύτερο να καλέσουμε για ακρόαση στην Επιτροπή μας το Διευθυντή, τον επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Κύριε Σεγητά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. θα μπορούσαμε ίσως να ακούσουμε τον ναι, που είναι ο εσωτερικό ελεγκτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οικονομικό ελεγκτή αρμόδιο για του οργανισμού, agencies. Obviously, the IAS is not responsible for taking disciplinary measures either. What we are Ούτε εμεί είμαστε υπεύθυνοι για την επιβολή κυρώσεων. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Κοιτάξαμε λοιπόν τα προγράμματα δράσης που μας υπέβαλε ο οργανισμός για να ανταποκριθεί στις συστάσεις της αρχής απαλλαγής όταν εσείς αποφασίσατε να αναβάλλετε την απαλλαγή. Και επίσης κοιτάξαμε και τα προγράμματα δράσης να, κατά πόσο να ακολουθούν τις δικές μας συστάσεις. Έτσι λοιπόν θεωρούμε, τουλάχιστον κατά την άποψή μας, λίγο πολύ ακολουθούν τις συστάσεις που και εμείς διατυπώσαμε και το Κοινοβούλιο, τα προγράμματα αυτά δράσης. Βέβαια το να υλοποιηθεί και κάθε συγκεκριμένο ένα πρόγραμμα δράσης είναι μια μεγάλη πρόκληση από μόνο του ως εγχείρημα και στο παρελθόν ο οργανισμός δυσκολεύτηκε να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό για να υλοποιήσει και τα συστήματα ελέγχου που χρειάζονταν. Κάτι που θα δυσκολέψει ίσως τον νέο διευθυντή. Αναζητούμε στήριξη από που μπορούμε. Η κυρία Ματσέ μας μίλησε για τις ημέρες εκπαίδευσης που και αυτή την εβδομάδα προβλέπονται Πιστεύουμε ότι είναι ένας επικοδομητικός τρόπος για να ενημερώσουμε το προσωπικό μας για το τι αναμένουμε σε σχέση με τους κανονισμούς της Επιτροπής. Επίσης, αργότερα φέτος, θα έχουμε μια ενημέρωση, όπως λέγεται, GAP για την υλοποίηση των εσωτερικών προδιαγραφών ελέγχου. Θα δούμε δηλαδή τι έχει υλοποιηθεί και τι απαιτείται βάσει αυτών των προδιαγραφών και θα διεξαγάγουμε και ελέγχους Ελέγχου παρακολούθησης για να δούμε τα προγράμματα δράσης έχουν όντω υλοποιηθεί και αν είναι αποτελεσματικά στην υλοποίηση, εάν πέτυχαν δηλαδή τους στόχου που είχαν τεθεί αρχικά. Ένας τέτοιος έλεγχος θα ξεκινήσει φέτος τον Οκτώβριο όπου θα κοιτάξουμε τον προγραμματισμό και το δημοσιονομικό σχεδιασμό των βασικών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και μαθημάτων και εκπαίδευση και θα δούμε πώ έχει προγραμματιστεί ο προπολογισμό του χρόνου. Θα δούμε πώ θα έχουν όλα αυτά διεξαχθεί, πώς θα έχουν υλοποιηθεί όλε οι δραστηριότητε του οργανισμού. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη φάση ο ρόλο μας είναι συμβουλευτικός και σε μια δεύτερη φάση πηγαίνουμε και ελέγχουμε κατά πόσο ακολουθήθηκαν οι συμβουλέ μα. Προεδρο ευχαριστούμε. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Σα θυμίζω ότι σε αντίθεση με όσα αναφέρει η μερίσια διαταξή, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 7η Σεπτεμβρίου και όχι η Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 8. Το πακέτο της εξωτερικής υπηρεσίας, διευθυντικός προπολογισμός 6-2010, τμήμα 2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τμήμα 10 Ευρωπαϊκή τμήμα 3 μάλλον Επιτροπή, τμήμα 10 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ο κύριος Μπαλτζήτη. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba e, nauja institucija. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση είναι νέο θεσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα νέο θεσμικό όργανο και πριν ιδρυθεί είχαμε πάρα πολλές άτυπες και επίσημες συνεδριάσεις και συζητήσεις. Εγώ είμαι συντάκτης νομοδότησης και έχω συντάξει την άποψή μου ε, και θα τη βρείτε και στο έγγραφο που σας έχω υποβάλει. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας αυτής η δημοσιονομική της ανεξαρτησία. Να προβλέπετε δηλαδή ξεχωριστό κεφάλαιο στον προπολογισμό. Συν το ότι θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς ο λειτουργικός από τον, τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει και ένα στοιχείο δημοσιονομικού ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου όμως για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και τις εξωτερικές δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα στη χορήγηση απαλλαγής και στην ΕΙΕΔ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όπως το πράττει αυτό το καιρό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να είναι ουδέτερη ε, η ε, κατάσταση αυτή, δηλαδή ουδέτερο ο προπολογισμό και να μην έχουμε επικαλύψει στη λειτουργία ούτε ε, στους πόρους από άλλες υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είναι επαρκής ε, και αποτελεσματική λειτουργία. Και βέβαια χρειάζεται εσωτερικό οικονομικό έλεγχο, Λογικό δεν είναι, άρα και επόμενο να προσαρμόσουμε τη γνωμοδότηση και να βεβαιωθούμε ότι ο εσωτερικός τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει και την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή ναι. Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Έχουν και την πραγματογνωμοσύνη και τα προσόντα. Οι ελεκτές Ευρωπαϊκή Επιτροπής γνωρίζουν ε, πώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, τι γίνεται με τι λειτουργικέ δαπάνε, τι γίνεται με τι επιχειρησιακέ δαπάνε, και θα είναι πιο εύκολο να κάνουν τον έλεγχο. Αφήστε δε που θα εξοικονομήσουμε και χρήματα σε αυτού του χαλεπού καιρού οικονομική ύφεση που διανύουμε. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής του δημοσιονομικού κανονισμού που ορίζει ότι ένα θεσμικό όργανο ε, θα κάνει το ίδιο τον εσωτερικό οικονομικό έλεγχο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους οργανισμούς. Εγώ θα πρότεινα να υπάρχει όχι μόνο μια υπηρεσία, αλλά ένας ελεγκτής που να ελέγχει και τις λειτουργικές δαπάνες και τις, και τις ε, επιχειρησιακές. Ναι. Και στο διοικητικό προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που προβλέπετε για τη λειτουργία από τους ιδίους πόρους θα ανηλυθούν αυτά τα κονδύλια ανάλογα με το ΕΠ του κάθε κράτους. 8,8 εκατομμύρια από τους ίδιους πόρους και τα υπόλοιπα από το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από χρήματα που πηγαίνουν στα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα λοιπά. Περίπου 600.000 από εκεί. Ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για την πρόσληψη προσωπικού, συντήρηση των κτηρίων και τις διοικητικές δαπάνες για το 2010. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δει κανεί αν είναι μεγάλη ή μικρή αύξηση του, ή πρικοδότηση του προπολογισμού. Δεν ξέρουμε. Νομίζουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερο να κρίνουμε μετά από ένα χρόνο λειτουργία του χρόνου τέτοιο καιρό, όταν θα ξέρουμε περίπου πώ θα έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια στου διαφόρου τομεί πολιτική. για να βγάλουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Και τώρα εκπρόσωπο τη Επιτροπή, εφόσον θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να εκχωρεί απαλλαγή για την υλοποίηση του συνόλου του προπολογισμού της Ένωσης δεν πλήττεται, ούτε μπορεί να πληγεί από το δευτερογενές δίκαιο ή από τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων. Αφού το έχουμε εξηγήσει αυτό, πρέπει να όμως να λάβουμε υπόψη βεβαίω και την ετήσια έκθεση δράσεων του δικαστηρίου που καλύπτει κάθε θεσμικό όργανο ξεχωριστά και τη διαχείριση του κάθε οργάνου. Και βάσει των ε, καθιερωμένων πρακτικών, το Κοινοβούλιο εξετάζει την υλοποίηση κάθε τμήματος του προπολογισμού, κάθε θεσμικού οργάνου ξεχωριστά Αυτό σημαίνει ότι ο προπολογισμό τη ΕΕ θα είναι πλέον θεσμικού οργάνου και θα είναι διοικητικό που θα περιέχει διοικητικέ ε, πιστώσει. Οπότε θα είναι υπεύθυνη η ΕΕ για την ε, υλοποίηση, την εκτέλεση του δικού της διοικητικού προπολογισμού. Και αυτό θα αποτελεί μέρος της διαδικασίας που θα ελέγξει και θα πρέπει να εκχωρήσει την απαλλαγή για αυτήν το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θα εκτελεί τον προπολογισμό, ιδίω ό,τι αφορά τι λειτουργικέ πιστώσει που βρίσκονται στο δικό του τμήμα, αυτό που του αναλογεί στον προπολογισμό και μόνο σε αυτό. Βεβαίω, η υλοποίηση αυτή των λειτουργικών πιστώσεων από την Επιτροπή ανέκαθεν αποτελούσε μέρο τη απαλλαγή που ελέγχει το Κοινοβούλιο. Πού εκχωρεί το Κοινοβούλιο. Συμπερασματικά λοιπόν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να εκχωρεί απαλλαγή παραμένει αναλύωτο. Δεν αλλάζει σε τίποτε από την δημιουργία της ΕΙΕΚ ως ξεχωριστού θεσμικού οργάνου και βάσει αυτού του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Ευχαριστούμε κυρία Γκρέσλη. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον πάντα να τα ακούει κανείς αυτά. Ε, περιμένω με χαρά την πρώτη απαλλαγή της ΕΕΔ και ε, de facto δεν είναι εύκολο να δώσουμε απαλλαγή σε ένα όργανο που δεν απορροφά το προϋπολογισμό του. Έτσι δεν είναι. Τελικά η πρέσβης, ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο εξωτερικό θα είναι αρμόδιος. Καλά και το οικοδόμημα έτσι κι είναι τελείως ε, ιδιάζων. Ε, θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε ε, κάπως λειτουργικό. Το θέμα είναι να σφίξουν τα πράγματα τι θα γίνει. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον. Ποιος θα μπορέσει να αποδείξει τι, αν χρειαστεί να το αποδείξει. Και εκεί κερδίζουν δύο η Υπηρεσία εξωτερική δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο χαμένος είναι ο φορολογούμενο που έτσι κι αλλιώ έχει συνηθίσει να είναι χαμένος τη υπόθεση. Είναι πολύ διχασμένα τα πνεύματα για το οικοδόμημα αυτό γιατί δεν είναι ούτε διαφανές και de facto ε, προκειμένου έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και δυσκολίες όχι μόνο εμείς αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσω στο σχέδιό μου για το δημοσιονομικό κανονισμό να το συγκεκριμενοποιήσω όσο γίνεται περισσότερο και στην πράξη να φέρω τον καθέναν ενώπιον των ευθυνών του. Για να μην αμφιβάλλετε καθόλου για τη φιλοδοξία μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί το ωραίο στην εξωτερική βοήθεια είναι ότι κάθε μέρα κάτι τρέχει κάπου. Δεν είναι κανένα τομέα που να δρανεί, α πούμε. Κάθε μέρα και από κάτι έχουμε. Το Αφγανιστάν είχαμε την περασμένη φορά και τα επόμενα έτη όχι μόνο στο Αφγανιστάν, Εντάσει θα έχουμε και στο Ιράκ, εμπόλεμε καταστάσεις, Γάζα, ξέρω εγώ, κοσφοπέδιο, δυσκολίες στον κόσμο και να είστε βέβαιοι ότι κάθε μέρα κάτι θα προκύπτει, κάπου συμβαίνει κάτι κάθε μέρα στον κόσμο. και αν γίνονται σφάλματα, προφανώ δεν εννοώ ότι φταίει κανένα για του πολέμου, αλλά αν γίνονται σφάλματα στη διαχείριση να δούμε πού θα βρούμε τον υπεύθυνο. Ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τον κύριο Παλτσίτη για την περασμένη εβδομάδα και τη συζήτηση και χαίρομαι πολύ. Και θα ήθελα να αξιοποιήσουμε όχι μόνο τον εσωτερικό ελεγκτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το λογιστήριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην έχουμε αλληλοκάλυψη, έτσι ε, διπλές δομές. Γιατί μόνο έτσι αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν θα είναι ε, μια κεντρική διοίκηση με διάφορα παραρτήματα διεθνώς. Γιατί αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Να, στήσουμε μια τεράστια μηχανή στην Κομισιόν με περισσότερες δαπάνες για τη διαχείριση κτλ. παρά για την εξωτερική βοήθεια. Θα πρέπει να είναι πολύ μικρή η διοίκηση και θα είναι και άτυπη η συμπεριφορά της σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υπόλοιπη. Και όποιος πάει εκεί στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα έχει σταδιοδρομία ε, πολύ ταχύτερη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιπτώσεις στους υπαλλήλου. Ερώτηση τώρα, τι γνωρίζουμε για το πόσο πάει το κόστος ε, των ε, διοικητικών δαπανών. Γιατί όποιον ρωτήσω μου λέει και άλλο αριθμό. Πόσο κοστίζει το χρόνο σε διοικητικέ. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν μπορούμε τώρα να το υπολογίσουμε, αλλά πώ το σχεδιάζεται για το 2011 ο διοικητικό προπολογισμό που καταρτίζεται, ποιο είναι, εκτό από τα επιπρόσθετα έξοδα. Εντάξει, μέχρι τρει μήνε. 10 εκατομμύρια ευρώ αυτά που είπατε για τρει μήνε, δηλαδή 40 το έτο. Πώ πάει αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προγραμματίζετε. Ευχαριστώ. Πρέγω. Παρακαλώ. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο κυρία Γκέσλερ. Για τρεις μήνες είναι τα 9 εκατομμύρια και για το 2011 το ποσό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το συζητάει ακόμη η Κομισιόν. Τις επόμενες μέρες, εβδομάδες θα το δούμε. Και περιμένει ακόμα η Κομισιόν να δει τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό. Σήμερα βέβαια δεν, είναι, δεν πρόκειται ακόμη για ενεργή δομή και έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να εξετάσει και να κάνει και κριτική αχρειαστή για τον προϋπολογισμό της ΕΑΕΣ. Κάνουμε όμως τα πράγματα, τα εξετάζουμε με την ίδια αυστηρότητα που κάνει και η Κομισιόν. Εγώ και οι συνάδελφοί μου κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε την ίδια δουλειά και δωρεάν για την ΕΑΕΣ εφόσον το δέχεται βέβαια, γιατί πρέπει το κάθε όργανο να καθορίσει και τον ταμεία του. Λογιστή. Η ε, κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ. Έχω και άλλες ερωτήσεις, ξέρετε, μου επιτρέπετε. Το παράρτημα 10 στον ε, κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τους εργαζομένους στις τρίτες χώρες αλλάζει επίσης. Ευχαριστώ για την πλήρη αδιαφάνεια εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Έχουμε συμβασιούχους που δεν έχουν τη ίδια μεταχειρίση με τους προσωρινούς υπαλλήλους ή τους μονίμους υπαλλήλους. Έχουμε διάφορες συμβάσεις και οι συμβασιούχοι δεν έχουν ας πούμε επιπλωμένα διαμερίσματα που δίνουμε στους προσωρινούς και στους μονίμους. Λοιπόν τώρα τους δίνουμε και διαμερίσματα και λέτε ότι δημοσιονομικά αυτό είναι ουδέτερο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό. Και ας πούμε, κλιματιστικά και συντήρηση. Μέχρι τώρα οι συμβασιούχοι τα πλήρωναν από την τσέπη τους. Και στη νέα υπηρεσία, στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ε, αυτοί ευθυγραμμίζονται με τους μονίμους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, de facto, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση καταργούμε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουμε καταλάβει αυτό και είναι ουδέτερο από πλευρά προπολογισμού. Δεν έχει επιπλέον κόστο. Υποθέτω ότι αυτά τα μικροκόστη θα χαθούν στο τεράστιο πακέτο, αλλά ε, θα ήταν δίκαιο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, τα μιλάμε για προπολογισμό, να πούμε τι σημαίνει αυτό. Όταν ευθυγραμμίζονται και ε, συστοιχίζονται, εν πάση περιπτώσει, οι συμβασιούχοι με τους υπολείπους ε, υπαλλήλους μας. Ευχαριστώ. Ε, thank ε, you Σας ευχαριστώ. Τις λεπτομέρειες για τα οικονομικά τις βλέπετε συνημένες στην πρότασή μας τροποποίηση του κανονισμού του προσωπικού. Η δυνατότητα λοιπόν των συμβασιούχων να παραμείνουν υπάρχει γιατί καμιά φορά έχουμε κενά τμήματα χωρίς υπαλλήλου. Κενά διαμερίσματα που δεν τα έχει καταλάβει κανένας υπάλληλος και μπορούμε να τα δώσουμε σε κάποιον συμβασιούχο. Η διαχείριση λοιπόν να γίνεται λίγο πιο ευέλικτα αντί να αρνούμαστε σε κάποιον συμβασιούχο το διαμέρισμα απλώς και μόνο γιατί είναι συμβασιούχος. Αν υπάρχουν κενά διαμερίσματα, τότε εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε τον νίκη και δεν είναι πρόσθετο κόστος αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. για τον προϋπολογισμό και αυτά που ακούσαμε τώρα. Και κατά πόσο συμβαδίζει με αυτά που έχουμε πει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι προϋπολογισμό θα έχουμε το 11, αλλά είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι προϋπολογισμό θα έχει η ΕΑΣ και για το 12 ακόμα. Γιατί διότι δεν μπορούν τα ποσά που έχουμε συζητήσει να πολλαπλασιαστούν κατά 3 και 4 διότι η ΕΑΣ θα έχει 1614 11 από την Κομισιόν και μόνο 100 καινούριου υπαλλήλου. Οι τρεις μήνες αυτοί θα χρηματοδοτηθούν από την Κομισιόν. Άρα ο προϋπολογισμός για τους μισθούς θα είναι τεράστιος και πολύ μεγαλύτερος από 40 εκατομμύρια. Και τα 9,5 εκατομμύρια διατίθενται για ενίκεια κτηρίων και γραφείων η δε προπολογισμός του 11 θα έχει και άλλο τρέχον κόστος που πρέπει από σήμερα να το δούμε. Η βασική ιδέα είναι ο διαχωρισμός ενός μέρους αυτού από την Κομισιόν να είναι πολύ σαφέστερος στο μέλλον για να ξέρουμε τι ακριβώς κάνει και πόσο κοστίζει η πρόταση αυτή να χρησιμοποιηθεί υπάρχουσα εμπειρία της Κομισιόν για τους λογαριασμούς είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να το λέει και η γνωμοδότηση. Το κυριότερο όμως είναι ότι πρέπει να περιμένουμε πότε θα μας έρθουν οι αναφορές, οι εκθέσεις για το κόστος που θα, για, τα κόστη που θα έχουν δαπανηθεί. Όχι μόνο για να γνωμοδοτήσουμε καλύτερα, αλλά και για να καταλάβουμε καλύτερα ποιος ακριβώς είναι, ποιο ακριβώς είναι το εύρος της εξωτερικής δράσης της Ένωσης ε, σε χώρες όπως το Αφιγανιστάν και άλλα, θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα και θέματα που δεν τα θίξαμε σήμερα καθόλου. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα περάσουμε στο σημείο 9. Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των κοινοτήτων. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Θα δώσω το λόγο στην ισχύτητα την κυρία Έρτσοκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο συντομότερα κινητά. Ε, θα προσέξουμε ιδιαίτερα ώστε ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο κανονισμός των υπαλλήλων να συμφωνεί με τις νομισμένες διαδικασίες, άρα να συμβάλλει και το Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα υποβάλει τη γνωμοδότησή της και σε άλλες επιτροπές με εισηγητή τον κύριο Μπένετ Τράμπκαη από την από την νομική. Για μένα το σημαντικότερο είναι να βρούμε έναν κάποιο μόντους βιβέντη για την υπηρεσία αυτή διότι το προσωπικό προέρχεται από τουλάχιστον τρία, τρεις πηγές την ίδια την Ένωση και τοπικά ειδικά συμβόλαια και η κυρία Γκλέσλερ θα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να υπάρξει διαμάχη συμφερόντων ιδιαίτερα για τους υπαλλήλους από τα κράτη-μέλη και από τα τοπικά συμβόλαια. Να μην υπάρχει διαμάχη συμφερόντων και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κανένα νέο συμβόλαιο δεν μπορεί να δοθεί σε προερχόμενο από χώρα που έχει ήδη χορηγήσει υπαλλήλους. Τώρα, οι υπάλληλοι από τα κράτη-μέλη και τα όργανα της Ένωσης. Εδώ πρέπει να λύθουμε ορισμένα προβλήματα. Πρώτα για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν ποιος θα διοριστεί και σε ποια θέση στο διπλωματικό σώμα. Αλλά Προς το παρόν έχουμε πει ότι θέλουμε και κάποιο είδους μετεκπαίδευση ώστε να γνωρίζουν όλοι τα ίδια πράγματα. Γιατί είναι βασικό αυτό αφού μιλάμε για προσόντα και Δεύτερον, η κινητικότης. Το 4 συν 4 που λέμε σε σύγκριση με την πενταετή θητεία των ευρωεπομπλατών, σημαίνει ότι αυτές οι διαφορές θα φανούν και στο κόστος μεταξύ των ειδών του προσωπικού. Άλλο σημαντικό θέμα. Οι διπλωμάτε που θα εργάζονται για την, εξωτερική, για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων θα έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα και ευθύνες και πρέπει επειδή αυτά θα καθοριστούν αργότερα όπως και η απαλλαγή μπορεί να έχουν επιστρέψει εντωμεταξύ στο κράτος τους. Αλλά η ευθύνη τους θα παραμείνει εδώ ακόμη και αν έχουν επιστρέψει. Εδώ. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα για μας από την Κοκομπού. Διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τελικές ευθύνες και οι δημοσιονομικές θα είναι σαφείς για οποιονδήποτε έρχεται από οποιαδήποτε υπαλληλική πηγή. Αυτό ήθελα να σας πω. Το έχω συζητήσει πολλές φορές με συναδέλφους, με τους σκιώδεις δηλαδή, και νομίζω ότι μπορούμε να τελειώσουμε τη δουλειά μας εν καιρό το δέοντι και εν ευθέτω χρόνο του, Ευαγγελίου, του της κοιμήσεως της Θεοτόκου λίγη διορία κατάθεσης των τροπολογιών. Ευχαριστούμε και τώρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή, εφόσον θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κανονισμοί εσωτερικής κατάστασης, όπως βλέπετε, περιέχονται σε ένα νέο έγγραφο και ήδη υπάρχουν διατάξεις σχετικές διότι οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τελείως άγνωστες. Έχουμε κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης για τα θεσμικά όργανα. Επίσης έχουμε κάποια ζητήματα σύγκρουσης φερόντων κάποιες φορές. Γι' αυτό υπάρχει ο τίτλο 2. Εκεί, στην κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ορίζονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων και των άλλων εργαζομένων. Εδώ μιλάμε επίση για ευθύνη και υπόλογο και υπάρχουν διατάξει που ισχύουν λόγω χάρη. Το άρθρο 22 του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση που θεωρούμε ότι αρκεί για να καλύψει οι καταστάσεις που μπορεί να ανακύψουν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτές οι διατάξεις δεν θα θέλαμε να επαναληφθούν και σε άλλα κεφάλαια κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και να ακολουθήσουμε μια συστηματική προσέγγιση σε όλα τα έγγραφα. Παρακαλώ, κύριε Γκρέσλε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τοπική είναι 3.000 οι ντόπιοι υπάλληλοι. Και δεν υπόκεινται στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων με τους υπολείπους. Και υπάρχουν και κάποια που εφαρμόζονται στους λοιπούς υπαλλήλους. Ε, αυτό δεν θα πρέπει να ισχύσει, το θεωρώ απολύτως απαραίτητο. Ευχαριστούμε. Όταν μιλούμε για λοιπούς εργαζομένους ή υπαλλήλους της Ένωσης, έχουμε τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης με τους ε, όρους πρόσληψης. Όμως, ο κανονισμός αυτός ισχύει κατά αναλογία και για άλλους εργαζομένους. Κατά αναλογία λοιπόν και για τους προσωρινούς ή για τους συμβασιούχους. Εάν κοιτάξετε το άρθρο 11 των όρων εργασίας, γίνεται αναφορά στον τίτλο 2 και δεν υπάρχει διαφορά στην μεταχείριση των υπαλλήλων και των προσωρινών συμβασιούχων εργαζομένων. Δεν ισχύει αυτό, δεν είναι σωστό, διότι μέχρι τώρα το γράφατε στις συμβάσεις εργασίας. Αλλά τι θα γίνει με τις 3.000 συμβάσεις για τους εγχώριους υπαλλήλους. Χρειάζεται να λυθεί αυτό. Το άρθρο 16 με 29 του ε, κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης δεν ισχύει για τους ντόπιου υπαλλήλους και θα πρέπει επιγόντως να τροποποιηθεί. Ευχαριστούμε. Μήπως θέλει η Επιτροπή και πάλι να παρέμβει. Κοιτάξτε, αν σωστά καταλαβαίνω, μιλάτε εσείς για τους τοπικούς και για αυτούς τους όρους εργασίας που ισχύουν για εκείνους. Όμως η ιδιαιτερότητα αυτών των τοπικών υπαλλήλων είναι ότι ενώ αναφέρονται στους όρους εργασίες, οι δικοί τους όροι εργασίες, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, δεν ορίζονται στους όρους εργασίας αυτούς καθεαυτούς. Διθετώνται από την εθνική νομοθεσία, εκεί ρυθμίζονται και αυτή υπερισχύει. Εάν υπάρχουν λοιπόν προβλήματα με αυτού του εργαζομένου, αυτού του υπαλλήλου, θα πρέπει κανεί να τρέξει στι εθνικέ δικαστικέ αρχέ και αστυνομικέ αρχέ για να επιλύσουν τα προβλήματά του. Ε, είναι λοιπόν κάπως διαφορετική περίπτωση. Διαφορετικό το πεδίο. Λοιπόν, η κυρία Γκρέσλε, σα σκέφη στο Αφγανιστάν και τις άλλες ε, ε, τέτοιες χώρες. Καλή τύχη. Θα πρέπει οι εντόπιοι υπάλληλοι να έχουν την ίδια μεταχείριση ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων πόθεν έσχεση για, ε, που ισχύει μάλλον και για τους ε, υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν αντιστοιχίες. Πάνε οι σύζυγοί τους και ανοίγουν εταιρείε και παίρνουν ε, προμήθειες και έργα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρουση συμφερόντων, εντάξει, επειδή είναι ντόπιοι. Πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Το βλέπω τελείω διαφορετικά. Και δεν μπορεί να παραμείνει αυτή η κατάσταση θεωρούσα ότι υπήρχε μια στοιχειώδη συνένεση για το τι απαιτούμε από τους υπαλλήλους μας. κατελάχιστο Με το αυτονόητο συζητάμε. Ευχαριστούμε εισηγήτρια. Νομίζω ότι είναι μείζονο σημασία το θέμα αυτό. Η ΕΕΔ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, να, δράσει, να ενεργεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Και μια από τι διαδικασίε αυτές θα είναι η διαδικασία απαλλαγή για να επιληφθούμε αυτού του θέματος. Έτσι λοιπόν συστήνω εντόνω, αν μπορώ να κάνω συστάση προς το Συμβούλιο, να κοιτάξει τις εκθέσεις απαλλαγή που κάναμε για την ε, υπηρεσία αναδιάρθρωση των Βαλκανίων και να κοιτάξω τα διδάγματα από εκείνη την εμπειρία. Διότι είδαμε περιπτώσεις το πώς μπορούν να δαπανώνται τα κονδύλια με αυτήν την υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν την διαδικασία αυτή που μαζί σχεδιάσαμε ως Επιτροπή σε σχέση με αυτόν τον οργανισμό να την ε, χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα και το δίδαγμα αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και για την ΕΕΔ για να αποσοβήσουμε τι ενδεχόμενε συγκρούσει συμφερόντων που μπορούν να συμβούν σε πολύ δύσκολε περιπτώσει και σε δύσκολε συνθήκε σε χώρε όπου το επίπεδο διαφθορά μπορεί να είναι υψηλό. Και πολύ μάλιστα υψηλότερο από ό,τι θα περίμενε κανεί για χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω τώρα. Άρα είναι σημαντικό σε ένα-δύο χρόνια να μην χρειαστεί να δούμε ποια τα λάθη που θα έχουμε κάνει τότε και να είναι αργά, να πρώτη τότε να τα διορθώσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αναδιάρθρωση των Βρετανίων ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό ω παράδειγμα για την ΕΕΒ και για το μέλλον. Σα ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Ε, Τώρα τα σημεία 10, 11 και 12 της εμερήσιας διάταξης, όπως είπα και στην αρχή, θα εξεταστούν αύριο από κοινού στην συνεδρίασή μας με την Επιτροπή Προεπολογισμών. Και τώρα έχουμε το σημείο 12.1. Διαθεσμική συμφωνία για συνεργασία σε θέματα οικονομικά και δημοσιονομικά. Εδώ θα σα κάνω μια σύντομη ανασκόπηση του θέματο, καθότι είμαι εγώ εισηγητή. Μετά τη συνεδρίαση, την κοινή συνεδρίαση τη 3η Μαρτίου, ορίστηκε εισηγητή για γνωμοδότηση που θα που ανέλαβε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και σε ό,τι αφορά τη διοργανική συμφωνία. Η διοργανική συμφωνία, όπως γνωρίζετε, μεταξύ Συμβουλίου Επιτροπής και Κοινοβουλίου για την συνεργασία στα δημοσιονομικά ζητήματα είναι μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των θεσμών που έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του προπολογισμού και είχε ως τώρα στα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε εδώ και για πρακτικές διευθετήσεις ό,τι αφορά το σύστημα του προπολογισμού, το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα και τα ανώτατα όρια και κατώτατα όρια του όλου προγραμματισμού. Η διοργανική συμφωνία, η προηγούμενη, διαφέρει από την τωρινή, καθότι τώρα το περιεχόμενο τη ισχύουσα συμφωνία μετά την ε, θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα θα παραπέμπει σε άλλε διαδικασίε. Έτσι λοιπόν για το πλαίσιο, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις ρυθμίσεις που είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο του τωρινού κειμένου, όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που ορίζει πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα για τα έτη 2007-2013. Άλλα τμήματα θα, θα συμπεριληφθούν μάλλον στις προτάσεις κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που θα τροποποιούν τον κανονισμό του Συμβουλίου 16, μάλλον, ναι, 1605 κάθετος 2002 για τον δημοσιονομικό κανονισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι η διαθεσμική συμφωνία αναφέρεται στις ρυθμίσεις της ε, ήδη υπάρχουσας συμφωνίας που δεν ε, καλύπτονται από τις δύο προτάσεις που σας προανέφερα. Έτσι, η Διοργανική Συμφωνία διέται σε τρίτα, τρία κεφάλαια. Η πρώτη αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο και τα συγκεκριμένα όργανα. Έπειτα το δεύτερο μέρο, η βελτίωση τη συνεργασία τη διαθεσμική στα πλαίσια τη διαδικασία του προπολογισμού. Και το τρίτο τμήμα αφορά την οικονομική διαχείριση των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο τμήμα παρουσιάζει τις γενικές αρχές που αφορούν την ε, διαχείριση δημοσιονομική. Η έκφραση αυτή, ο όρος όπως χρησιμοποιείται στο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας, περιορίζεται σε τρία ζητήματα που καλύπτονται σε τρία υποκεφάλαια. Δημοσιονομικός προγραμματισμός, ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και δημοσιονομικοί μηχανισμοί, εργαλεία. Έτσι λοιπόν δεν βρισκόμαστε εδώ στο κατάλληλο πλαίσιο για να υποβάλουμε διεξοδικέ προτάσει για την εξυγίανση και την προγραμματισμό του, δημοσιονομικού μας, του νέου δημοσιονομικού προγραμματισμού. Αυτό θα γίνει με τον τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου και την ενδεχόμενη εξέταση του σχεδίου προπολογισμού στην φυσική έδρα όπου πρέπει να εξεταστεί το θέμα, το, θέμα αυτό. Έτσι δεν θα επικαλύπτονται οι πολυάριθμες διαδικασίες που αυτή τη στιγμή βρισκόνται σε εξέλιξη και σε διαπραγμάτευση. Γι' αυτό η γνωμοδότησή μα θα παραμείνει στα σημεία τη Διόργανική Συμφωνία, που αφορούν συγκεκριμένα τι αρχέ που εφάπτονται των ζητημάτων τη δική μα επιτροπή. Και τα υπόλοιπα σημεία του δημοσιονομικού κανονισμού θα καλυφθούν, όπω σα είπα, από την άλλη Επιτροπή. Έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο για τα νέα δημοσιονομικά μέσα. Το σχέδιο Διοργανική συμφωνία περιλαμβάνει την εξή έκφραση που θα το εξή ε, κείμενο που διαβάζω. Οι μηχανισμοί χρηματοδότηση και οι μηχανισμοί συγχρηματοδότηση χρειάζονται για να ενισχύσουν την ε, αυξητική τάση του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντα περισσότερα κίνητρα για χρηματοδοτήσει. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δημοσιονομικών μέσων, πολιετών και τέτοιου είδου που να δράσουν ως ε, καταλήτες για δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσεις. Τη στιγμή υποβολής του σχεδίου προπολογισμού η Επιτροπή αναφέρεται στις δημοσιονομικές αρχές για τις δράσεις που έχουν ε, χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναδιάρθρωσης για την ανάπτυξη και την στήριξη των ε, ε, δράσεων της ε, έρευνας και της ανάπτυξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δημοσιονομικά μέσα, τα πολιετή δημοσιονομικά μέσα πρέπει να δρουν ως καταλήτες για τους ιδιώτες επενδυτές και δημόσιους επενδυτές και για την δημιουργία σχέσεων εταιρικών ε, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έπειτα, για τον δημοσιονομικό έλεγχο, το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και εδώ καλό θα ήταν να έχουμε περισσότερα στοιχεία και από την πλευρά της Επιτροπής, ιδίως για το θέμα ότι οι φορείς αυτοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους αρχές της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Δεν αρκεί να λέμε ότι οι αρχές αυτές είναι επαρκείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την πρόταση δημοσιονομικού κανονισμού, εντοπίζουμε στην πρόταση της τριετούς αναδιατύπωσης του κανονισμού ότι η Επιτροπή θέλει να διευκολύνει την ευρύτερη ε, χρήση των ε, δημόσιων εταιρικών ε, σχέσεων. Εδώ βάσει του άρθρου 185 και 108 κυρίως. Προτείνονται έτσι από τη μια η ανάθεση εκτέλεσης μεικτών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών δράσεων, δημόσιων και ιδιωτικών και η χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια, λόγου χάρη με την ε, διαδικασία ανάθεσης και με την έμεση χρηματοδότηση. Έτσι με τις εκχωρούμενες αρμοδιότητες προβλέπεται ένα ελαφρύ σχέδιο προπολογισμού το οποίο θα επιτρέψει τη δημιουργία ακριβώς τέτοιων μεικτών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή λοιπόν υποβάλλει εδώ την ευρύτερη χρήση των ε, επιχειρηματικών αυτών ε, μορφών και προάγει την ευρύτερη ακριβώς ε, χρήση τους. Οι δημόσιες ιδιωτικές όμως αυτές οι επιχειρηματικές δράσεις δεν είναι ο μονός τρόπος για να επιτευχθούν οι πολιτικοί στόχοι που έχουν τεθεί. <clears throat> Απλώς είναι ένα καλό κίνητρο και μια καλή ευκαιρία αυτή για να εξερκίσουμε γιατί αυτοί οι μεικτές, οι κοινέ ε, δράσεις είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Το δεύτερο σημείο που μας απασχολεί και απασχολεί τον εισηγητή είναι η αδυναμία της αναφοράς στην απουσία συγκεκριμένων ετοιμάτων ελέγχου ό,τι αφορά αυτέ τι μεικτέ επιχειρήσει ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Στην πραγματικότητα, το κείμενο που σα ανέφερα στα πλαίσια τη διοργανική συμφωνία και στο νέο σχέδιο κανονισμού και σε ό,τι αφορά τη σχέση της Επιτροπής με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας και τη διαδικασία προπολογισμού και την εξυγίανση ή τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Εκεί η Επιτροπή αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Ούτε διαβλέπει την ανάγκη αλλαγών. Στο σημείο αυτό εδώ εγώ τουλάχιστον διαβλέπω την ανάγκη να εξηγηθεί καλύτερα ο τρόπο λειτουργία των ε, μεικτών αυτών επιχειρήσεων ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να αναλυθούν ε, διεξοδικά και με ανοιχτό πνεύμα για να καταλάβουμε αν είναι ο βέλτιστο τρόπο για να, για να παρέχονται και δημόσιε υπηρεσίε και βάσει τις εμπειρία που έχουμε από Ευρωπαϊκέ χώρε ό,τι αφορά την διαχείριση των δημόσιων κονδυλίων από τι μεικτέ αυτέ επιχειρήσει. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τα ζητήματα τα λογιστικά ελέγχου και ευθύνη των σχέσεων του, δημο... του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό. Και όλα αυτά πρέπει να αποσαφινιστούν. Και είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εύρωστη και υγιή διαχείριση των μεικτών αυτών επιχειρήσεων, να υπάρχει πρόσβαση στο ενεκτικό συνέδριο και στην υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης Όλαφ και επίσης να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει συμμόρφωση των μεικτών αυτών επιχειρήσεων με το δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες του. Εκεί θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσουμε την συζήτησή μα και περιμένω εδώ τη συνεισφορά και τα σχόλια όλων των συναδέλφων. Στο πούντο Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν έτσι κάποιες διαδικασίες στο Κοινοβούλιο που είναι δυσάρεστε σε όλους τους συναδέλφους και όχι δημοφιλείς, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ακριβώς εκεί κρίνεται το αν θα κερδίσουμε ή αν θα χάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που αναλάβατε να μας ε, βγάλετε από τη δύσκολη κατάσταση, να δούμε τι κάνουμε με τα νέα χρηματοδοτικά ε, μέσα. Αυτά βγαίνουν σαν μανιτάρια, ξεφυτρώνουν συνέχεια και έχουν το εξής κοινό όλα. Σε τελική ανάλυση δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν έχουμε ούτε δικαίωμα λόγου, ούτε δικαίωμα ελέγχου, ούτε τίποτα άλλο, γιατί είναι επιπλέον δουλειά, δηλαδή πλήρης αδιαφάνεια και εδώ στα χρηματοδοτικά μέσα, έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να εκφράσω την κριτική μου ρητά και σε σχέση με τα όσα αποφάσισε το Κοινοβούλιο αυτό συμφωνεί. Στην έκθεση Λιμπεράτσκι και στην έκθεση ΟΝΤΗ για την απαλλαγή ε, ε, φράσαμε μεγάλες επικρίσεις γιατί λείπει και διαφάνεια και ε, ο λόγος του Κοινοβουλίου ότι περνάει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι στο δικό μας πεδίο και βάζουν χέρι στις δικές μας αρμοδιότητες. Πώς μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή να μεταφέρουμε εκεί δραστηριότητες. Θα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Γιατί τελικά δεν ελέγχει κανείς κανένα. Το είδαμε και στους οργανισμούς σήμερα ε, πού ε, πάει η κατάσταση, πώς ξυλώνεται ο δημόσιος έλεγχος και είναι λιγότερος δημόσιος έλεγχος στους οργανισμούς. Ε, γιατί ε, μας ξεφεύγει αυτό, διαφεύγει το ελέγχο μας και δεν είναι προς το συμφέρον μας να επεκταθούν αυτά τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά μέσα και να στέλνουμε λεφτά εκεί και να μην έχουμε κανένα έλεγχο. Να μην έχουμε κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο, ούτε να μπορούμε να εφαρμόζουμε ε, διάφορα μέτρα και για ένα στοιχειώδη έλεγχο θα πρέπει να αγωνιζόμαστε συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό να συνεχίζεται, καταστρέφουν ε, το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε ε, να τα βλέπουμε έτσι αυτά να συμβαίνουν ε, χωρίς αντίδραση. Να είμαστε λοιπόν επικριτικοί και να τα λέμε. Χάνουμε δικαιώματα εδώ και να σταματήσει. Αρκετά μας πήραν μέχρι εδώ. Ε, Σας ευχαριστώ κύριο Σοντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, νομίζω, όπως και η κυρία Γκρέσλε, πρέπει και εμείς να ασκήσουμε εδώ τα δικαιώματα ελέγχου, δημοσιονομικού ελέγχου που περιμένουν από εμά οι πολίτες, γιατί αυτό είναι το ίδιο κάθε κοινοβουλίου. Όπως είπατε πρόεδρε, για τα νέα δημοσιονομικά εργαλεία, τα νέα δημοσιονομικά μέσα έχουμε δεχτεί εδώ την υλοποίηση ενό πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Εδώ το έχουμε συζητήσει διαμακρό με την κυρία Πασό. Και νομίζω ότι εδώ η δομή του προπολογισμού θα πρέπει να επιτρέπει περισσότερες επενδύσεις. Αν κοιτάξει κανεί. τι έγινε με το Γαλιλαίο, με το Ίτερ. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα και από τεχνικής άποψης και δημοσιονομικής έχουμε δυσκολία να το ελέγξουμε. Έτσι, στη χώρα μου, λόγου χάρη, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν δικό τους τμήμα λειτουργίας και ένα ιδιαίτερο προπολογισμό για τις επενδύσεις. Υπάρχουν διαφορετικέ αρχέ για αυτά. Και εδώ λοιπόν θα έπρεπε να προβλέψουμε συγκεκριμένα μέσα και ταξινομήσει στον προπολογισμό ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε ει πέρα τέτοιε μεγάλε επιχειρήσει, ε, τέτοια μεγάλα εγχειρήματα πολιετή. Διότι πιστεύω ότι ένα μέρο των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο και σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Υπήρου για τις τεχνολογίες, για τις θαλάσσιες οδού, για τις ποτάμιες οδούς, για την τεχνολογία, την υγεία, το διάστημα. Υπάρχει ένα σύνολο μεγάλων προγραμμάτων και εγχειρημάτων για τα οποία θα είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι και να διαρθρώσουμε σωστά τον προπολογισμό μας και να μπορούμε και να τον ελέγξουμε. Εδώ κάπως διαφωνώ με όσα είπε η Ίγκε σε μερικά σημεία, αλλά σε γενικές γραμμές συμφωνώ με το γενικό της προσανατολισμό. Grazie, onorevole Συγγνώμη, ε, τώρα βρήκα το σημείωμά μου, έχω και άλλα να σας πω. Θα πρέπει να γράψουμε επίσης ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός προέχει από τις επιμέρους κλαδικές ρυθμίσεις. Έτσι, προέχει ο δημοσιονομικός κανονισμός από τους επιμέρους κανονισμούς του κάθε ταμείου. Να το προσθέσουμε αυτό, είναι σημαντικό. Και επίσης να κάνουμε και άλλο αυτοπεριορισμό των προγραμμάτων. Έτσι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο το 2011 η Συντονία Ζεζεύσκα, για πώς τη λένε αυτή, είναι η βασική συγγήτρια για τον προϋπολογισμό γενική και λέει πόσα λεφτά ε, έχουμε ε, για προγράμματα νεολαία. Έχουμε πάνω από 10 προγράμματα για τους νέους, με γελία ποσά στο καθένα και τελικά μια τρύπα στο νερό κάνουμε. Λοιπόν, να περιορίσουμε και τον αριθμό των προγραμμάτων. Καλύτερα λίγα και καλά, αλλά με σωστή χρηματοδότηση, με μεγάλο ειδικό βάρος, παρά να έχουμε πληθώρα προγραμμάτων. Το ίδιο ισχύει και αλλού για τους πολλούς κανόνες και τα πολλά προγράμματα. Και αυτά να τα περιορίσουμε. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή αν θέλει να παρέμβει. Πρόεδρε. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση κάλυψε διάφορα θέματα. Για του, τις δικαιοσύνες ελέγχου του Κοινοβουλίου καταρχάς όλα αυτά πρέπει να συμπληρωθούν από τον τρόπο εφαρμογής που δεν τα λέει αυτά ο κανονισμός. Ούτως ή άλλως στο 53β υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις, ιδιαίτερα ο εσωτερικός έλεγχος, και η αναγκαιότητα να υπάρξει ένας ανεξάρτητος δημοσιονομικός έλεγχος για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ούτως ή άλλως λοιπόν οι δικαιοδοσίες ελέγχου της αρχής του προϋπολογισμού θα τύχουν σεβασμού. Οι σχέσεις μας με την ΕΤΕ είναι απαραίτητες γιατί δεν έχουμε στην Κομισιόν όλη την τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε. Ήδη σημειώθηκαν επιτυχίες από τέτοια συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία και ελπίζω και από τον Ιερεμία να δείτε πόσο επιτυχή είναι όλα αυτά. Τώρα, για τη δυνατότητα δανειοληψίας από τις ε, συλλογικές, τοπικές αρχές μάλλον, εδώ χρειάζεται η ανάγκη πολυετούς σεβασμού υποχρεώσεων ενώ ο προπολογισμό έχει ενιάυσιο χαρακτήρα. Άρα εδώ χρειάζονται επενδύσεις, οι αιτήσιες δαπάνες επί μεγάλη σειρά ετών βέβαια μπορούν να αποτελέσουν μια επένδυση αλλά βέβαια διαφέρουν οι μηχανισμοί ανάλογα με τις τοπικές αρχές και εξαρτώνται όλα αυτά και από τη δυνατότητά τους να δανειολείψουν. Κυρία Γκρέσλερ, εγώ δεν είμαι βέβαιος και λυπάμαι γι' αυτό ότι δίνεται όντως προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα. Εδώ οι νομομαθείς μου λένε ότι δεν υπάρχει αναγκαστικά κάποια ιεράρχηση Αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε εμείς στην Κομισιόν και